Uh, uh, Καλημέρα σας. Θέλω να σας επαναφέρω όλους στην τάξη και να ξεκινήσουμε τη δεύτερη συνεδρίαση ε, της Επιτροπής μας αυτή την εβδομάδα και είμαι πανευτυχής ε, να ε, έχω εδώ τον καθηγητή Μάριο Μόντι για τη δεύτερη φορά εφέτος ο οποίος θα μας παρουσιάσει ορισμένες από τις ιδέες ε, τις οποίες επεξεργάζεται εις την έκθεση που καταρτίζει για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επανακίνηση της ενιαίας αγοράς. Ξέρετε ότι είναι ένα, ε, το θέμα μας τον απασχολεί πάρα πολύ και νομίζω ότι θα παρουσιάσει ορισμένες από τις ιδέες μας Στι στις μελλοντικές του εκθέσεις. Άρα με τα μεγάλης χαράς θα τον ακούσουμε όπως και τον κύριο Λουί Γκρέκ τον οποίο, στον οποίο θα δώσω το λόγο στη συνέχεια για να παρουσιάσει την πολύ ενδιαφέρουσα έκθεσή του και ε, θα έχουμε μία πρώτη ανταλλαγή ε, στις ε, απόψεων μετά θα έχουμε στις 10 ε, τις ψηφοφορίες και θα μπορέσει να πιει ένα καφέ ο καθηγητής Μόντι και στις 11 θα, όταν τελειώσουμε θα μας παρουσιάσει την ομιλία του και θα συζητήσουμε την έκθεση Γκρέκ και την έκθεση ε, Μόντι. Αυτό σε αυτό θα αφιερώσουμε ε, τις συζητήσεις μας ε, σήμερα για την ενία αγορά. Αυτά σας περιμένουν λοιπόν εδώ σήμερα και προτού ε, προχωρήσουμε έχω ένα βασικό θέμα να σας αναφέρω. Δηλαδή νομίζω ότι όλοι οι συνάδελφοι γνωρίζουν ότι τώρα πολύ σωστά κατά τη γνώμη μου πρέπει ε, να ε, διατυπώσουμε πιο επίσημα εάν οι εισηγητές της Επιτροπής θα πρέπει να καταλήγουν σε συζητήσεις πρώτης αναγνώρισης γνώσεως για εκθέσεις. Ε, τυπικά πρέπει να το αποδεχτούμε. Έχουμε ε, και την έκθεση της κυρίας Βάισμπεργκερ για την απόρριψη ορισμένων ε, νομοθετημάτων βάσει της Επιτροπολογίας. Η κυρία Βάισμπεργκερ ήρθε χθε να μας πει και μας είπε ότι θα έπρεπε να συνεχίσουμε τις συζητήσεις για την κατάληξη σε πρώτη ανάγνωση. Θα τους δώσω το λόγο στη συνέχεια και μετά θα σας υποβάλω την πρότασή της επισήμως για να συμφωνήσουμε αν ε, ε, πρέπει να συνεχίσουμε από αυτή τη βάση. Καταρχήν της δίνω το λόγο. Ευχαριστώ κύριε ε, Πρόεδρε. Και εγώ πιστεύω ότι σε αυτές τις πολύ τεχνικές εκθέσεις όπως πολύ σωστά είπε και η κυρία Γκέπχαρτ εχθές στις διαπραγματεύσεις για τον τριμερή διάλογο μπορούμε να προχωρήσουμε και Πιστεύω ότι σωστό είναι να ακολουθήσουμε αυτή την τυπική διαδικασία διότι ε, υπάρχουν ε, εντωμεταξύ ενημερώσεις για τον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται οι διαπραγματεύσεις. Με μία λοιπόν διαπραγμάτευση με τον τριμερή, σε τριμερή διάλογο μπορέσαμε να καταλήξουμε σε μία έκθεση και πιστεύω ότι ο σε ορισμένες περιπτώσεις δεν αξίζει να προχωρήσουμε στη δεύτερη ανάγνωση και ε, χθε ε, στη συνεδρίαση των συντονιστών ε, μου εδόθη η άδεια και σήμερα από τις 8 το πρωί χωρίς πρωινό συναντήθηκα με τους σκιώδεις εισηγητές για να μπορέσουμε να διαγράψουμε μία γραμμή γραμμή πλεύσεως σύμφωνα με αυτά που είπε η κυρία Γέφερτ και υπέβαλα μία πρόταση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να προχωρήσουμε στις διαπραγματεύσεις. Άρα σήμερα το απόγευμα έχουμε μία θέση έτοιμη για τον τριμερή διάλογο και γι' αυτό θα ήθελα να προτείνω στην Επιτροπή επειδή ο φάκελος είναι πάρα πολύ τεχνικός να συμφωνήσει. Θέλω βέβαια να ευχαριστήσω για την πολύ επικοδομητική συνεργασία με όλους τους συμμετέχοντες. Ήταν μια πολύ ευχάριστη εμπειρία. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκέπχαρτ. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Βάις Γκέρμπε ε, διότι συνεργαστήκαμε πάρα πολύ καλά ε, σχετικά με το θέμα αυτό και θα ήθελα και εδώ να επαναλάβω προτού λάβουμε μία απόφαση ότι εχθές το βράδυ στη συνεδρίαση των συντονιστών είπα κάτι που είναι πολύ βασικό για την πολιτική μου ομάδα. Δηλαδή εδώ είμαστε σήμερα έτοιμοι εξαιρετικά να δεχθούμε να υπάρξει μία κατάληξη σε πρώτη πρώτη ανάγνωση και αυτό δεν πρέπει επουδενή λόγο να αποτελέσει ένα προηγούμενο διότι η πολιτική μου ομάδα είναι της γνώμης ότι υπό μαλάς συνθήκας πρέπει να προχωρούμε στην διαδικασία δύο αναγνώσεων που πρέπει να διατηρηθούν διότι ε, αυτό έχει μεγάλη σημασία για τους πολίτες. Εδώ όμως ε, εξαιρετικά επειδή είναι πολύ τεχνική έκθεση και επειδή υπάρχει ευρεία συνένεση στο Κοινοβούλιο και ε, υπάρχει μια ευρεία συνένεση μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου επειδή ε, συγκλίνουν αυτές οι τρεις, ε, αυτά τα τρία θέματα γι' αυτό εξαιρετικά δέχομαι αυτή τη διαδικασία. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, μπορώ τότε να ε, προεξοφλήσω ότι δέχεστε τη θέση αυτή και ο πρώτος θερμιερής διάλογος θα είναι σήμερα το απόγευμα στη μία. Οπότε δεν θα χάσετε μόνο το πρωινό σας αλλά και το μεσημεριανό σας γεύμα. Δεύτερον, είχαμε μια πολύ επικοδομητική και μακρά συνάντηση συντονιστών εχθέ το βράδυ ε, και θέλω να τονίσω ορισμένα από τα συμπεφωνημένα. Ε, καταρχήν θα υπάρξει μια γνωμοδότηση για την Επιτροπή Αναφορών που αναφέρεται σε μια αναφορά και η οποία έχει ε, σταλεί από την Αυστραλία Αυστραλία για να απαγορευτεί η εισαγωγή δέρματος καγκορού προς την Ευρώπη. Ε, επίσης θέλουμε να υπάρξει μία ακρόαση για το μέλλον της ευρωπαϊκής τοπικής τυποποίησης τον Ιούνιο σχετικά με την έκθεση και για την τυποποίηση και προβλέπουμε και ένα εργαστήριο, ένα workshop για το μέλλον της ενιαίας αγοράς για να γίνει ένα ευρύτερο φόρουμ ενιαίας αγοράς ε, μαζί με εκδηλώσεις που προβλέπονται για το 2011. Αυτά, ε, ε, αυτές είναι πτυχές των της του ψηφίσματος ή των ψηφισμάτων που είχαμε ε, στο Στρασβούργο σχετικά με το Solvit και το πίνακα βαθμολόγησης της ενιαίας αγοράς. Ε, όσον αφορά τα υπόλοιπα θέματα μπορείτε να τα διαβάσετε εις, ε, τα πρακτικά της συνάντησης των συντονιστών όταν θα δημοσιευθούν. Άρα προχωρούμε στη σημερινή μας συνεδρίαση και καλωσορίζω και πάλι τον Αντιπρόεδρο Λουί που παρουσίασε μία πολύ ενδιαφέρουσα και προκλητική ε, έκθεση, σχέδιο εκθέσεως ουσιαστικά ε, για την ενιαία αγορά και μετά ε, θα δώσω τον λόγο εις τους πιο ηγητές, Ροσφόρ, Χάνβας, Διόν, ο κύριος Σαβινί δεν είναι εδώ αλλά φαντάζομαι ότι θα έρθει. βλέπω ότι και η εκπρόσωπος της Επιτροπής που είναι φίλη της Επιτροπής είναι ε, παρίσταται εδώ και έτσι τώρα προχωράμε στην πρώτη συνεδρίαση και δίνω το λόγο στον Λουί Γκρέκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα <clears throat> να καλωσορίσω τον καθηγητή Μόντι που είναι παρόν σήμερα για την ανταλλαγή απόψεων για την εσωτερική αγορά και την υλοποίησή της όπως γνωρίζετε. Ο καθηγητής ε, Μόντι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τον Πρόεδρο Βαρόζο είχε επιφορτιστεί με το ε, καθήκον να εξετάσει τις προοπτικές για την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς. Η δική, ε, η δική μου έκθεση είναι η αντίδραση της ΣΥΝΚΟ για την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς και εδώ έχει εμπλέκεται και το έργο του κυρίου Μόντι. Έχουμε εδώ τις απόψεις ε, για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της ε, εσωτερικής αγοράς όσον αφορά τους πολίτες και τους καταναλωτές. Πρόεδρε, από το 1992 η εσωτερική αγορά <clears throat> έζησε τρεις διευρύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης είδε την ανάδυση μεγάλων οικονομιών όπως της Κίνας και της Ινδίας και πιο πρόσφατα αντιμετώπισε την πιο σκληρή περίοδο κρίσης της ιστορίας της Ένωσης που απειλεί να διακυβεύσει την ε, ε, ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. Εν ώψη αυτού του σκηνικού συνέταξα εγώ την έκθεσή μου. Ουσιαστικά η έκθεσή μου στοχεύει να θεωρήσει την ε, Ευρωπαϊκή Ενιαία Εσωτερική Αγορά υπό μακροοικονομική πρόπτική, λαμβάνοντας υπόψη φυσικά το πλαίσιο του 2020, ε, τη στρατηγική για το 2020, καθώς και την πρόσφατη χρηματοοικονομική κρίση. Όπως καταδεικνύεται πρόσφατα από την κρίση στις χρηματοοικονομικές αγορές, δεν υπάρχουν δεδομένοι νόμοι μέσα στο οποίο το περιβάλλον το οποίο δημιουργείται για την εσωτερική αγορά να είναι δεδομένο. Υπάρχει ρευστό κατάσταση και ε, πολλές δυνάμεις που επηρεάζουν αυτήν την κατάσταση. Η εσωτερική αγορά όσον αφορά το προστατευτικό ε, κλίμα που ε, απορρέει από αυτή την κρίση γίνεται πολύ πιο ευάλωτη. Σαν συνέπεια τούτων θα πρέπει να πληρώσουμε το αντίτιμο της ε, υποβάθμισης ε, της ε, εκτίμησης και των αποτελεσμάτων αυτής της κρίσης στην εσωτερική αγορά. Όμως πιστεύω ότι μπορούμε να κερδίσουμε από το να ταυτοποιήσουμε τα λάθη από το παρελθόν, να μάθουμε ελπίζω τα μαθήματα από αυτά τα βιώματα και να συνεισφέρουμε ώστε να υπάρξει μια θετική αλλαγή και όχι τόσο να βασιζόμαστε σε μια αναποτελεσματική μεθοδολογία και στην τύχη. Μπορούμε να δημιουργήσουμε μια ευκαιρία από αυτή την κρίση, να αλλάξει η νοοτροπία των πολιτών, να αναζωογονήσουμε το σχέδιο της ενιαίας εσωτερικής αγοράς, ώστε να ξεφύγουμε από τα λιμνάζοντα ύδατα. Τούτων λεχθέντων όμως δεν θα πρέπει όλη η μελλοντική μας στρατηγική να βασίζεται στην βραχυπρόθεσμη διαχείριση και αντιμετώπιση της κρίσης επί σειρά ετών η ενιαία εσωτερική αγορά <clears throat> απέτυχε να πείσει τους Ευρωπαίους πολίτες ότι πραγματικά εκπροσωπεί τα συμφέροντά τους και τις φιλοδοξίες τους. Αυτό που είναι ακόμα πιο σημαντικό είναι οι πολίτες και οι καταναλωτές φυσικά να δούμε ότι όλο και περισσότερο αισθάνονται ανασφαλείς χάνουν την εμπιστοσύνη τους στις αγορές. Μια επαρκής γνώση λοιπόν των <clears throat> δικαιωμάτων τους μέσα στο πλαίσιο αυτό, μια πολύ περίπλοκη νομοθεσία σε συνδυασμό με μια μη ευδιάκριτη εικόνα της ενιαίας εσωτερικής αγοράς υπήρχαν ως αρνητικά στοιχεία πριν από την κρίση ήδη. Είναι σημαντικό λοιπόν να αναγνωρίσουμε ότι ο παραδοσιακός ορισμός της ενιαίας εσωτερικής αγοράς ότι δηλαδή συνδέεται μόνο αποκλειστικά στην οικονομική σφαίρα πρέπει να αναθεωρηθεί. Μια νέα ολιστική συνολική προσέγγιση πρέπει να εφαρμοστεί όσον αφορά τι αγορέ. Μια που να εντάσσει τι ανησυχίε και τα μελήματα των καταναλωτών δίνοντά του ε, κέριο ρόλο κεντρικού πρωταγωνιστή στην ε, λειτουργία τη εσωτερική αγορά. Η αναζωογόνηση λοιπόν τη ενιαία εσωτερική αγορά μπορεί να επιτευχθεί με μια πιο πειθαρχημένη προσέγγιση χωρί να περιοριζόμαστε υπερβολικά υπερβολικά από δογματισμούς και ιδεολογίες, ιδεολειψίες. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή η προσέγγιση θα πρέπει να ενσωματώνει τα οικονομικά, κοινωνικά και <clears throat> περιβαλλοντικά μελήματα και ανησυχίες των Ευρωπαίων καταναλωτών, πολιτών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Επίσης Θέλω να υπάρξει μια πραγματικά πράσινη εσωτερική αγορά, αναγνωρίζοντας ότι το διαδίκτυο, η έρευνα, η ανάπτυξη, η καινοτομία, η γνώση πρέπει να διαδραματίσουν ένα πολύ θετικό ρόλο για τη μελλοντική διαμόρφωση αυτής της εσωτερικής αγοράς. Είναι λοιπόν προφανές τούτων λεχθέντων ότι μια καλώ λειτουργούσα και ολοκληρωμένη εσωτερική αγορά είναι αναγκαία προπόθεση για να εμβαθυνθεί η ολοκλήρωση στην Ευρώπη. Κοινωνική συνοχή, οικονομική ανάπτυξη και αηφόρο ανάπτυξη όσον αφορά την Ευρώπη. Όλοι είμαστε επισμένοι. Τώρα επιτέλου είναι η χρονική στιγμή για δράση και ότι η ενιαία εσωτερική αγορά πραγματικά χρειάζεται κατεπηγόντω μια νέα όθηση, νέα κίνητρα. Υπάρχει ευρεία συνένεση ότι μια πραγματικά νέα ε, καθέλκυση της εσωτερικής αγοράς απαιτεί στοχοθετημένες στρατηγικές που θα είναι ολοκληρωμένες και επικοδομητικές και που θα δίνουν τα αναγκαία αυτά προτερήματα οικονομικά και ανταγωνιστικά διασφαλίζοντας ταυτόχρονα της κοινωνική, την κοινωνική διάσταση. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι μια νέα ατζέντα, μια νέα ημερήσια διάταξη για αυτή την εσωτερική αγορά δεν θα είναι υπερβολικά ευρεία και υπερφορτωμένη και σαν αποτέλεσμα αυτού κάθε αντικείμενο να είναι προτεραιότητα ένα σημαντικό μέσο είναι η σωστή επιλογή προτεραιοτήτων και η ιεράρχηση αυτών των προτεραιοτήτων για το μέλλον. Σε αυτή την έκθεση επίσης εξετάσαμε τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν ώστε να πετύχουμε μια πιο πλήρη ενιαία εσωτερική αγορά. Τούτων λοιπόν λεχθέντων ωστόσο από την άλλη πλευρά θεωρώ προσωπικά ότι σε αυτή τη χρονική στιγμή στην εσωτερική αγορά αντιμετωπίζουμε διαφορετικά προσκόμματα και θέματα και ξεκινώντας από προβλήματα νοοτροπίας Μπορούμε όμως να ανοίξουμε, αν δεν είμαστε ε, σταθεροί στην αντιμετώπιση των προκλήσεων, μία, ε, το πίθο των Δαναίδων. Γι' αυτό πρέπει να μην ε, υποεκτιμούμε τις προκλήσεις όσον αφορά τις διαφορετικές απόψεις και τις, το περίπλοκο πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να δράσουμε. Επίσης στην έκθεσή μου εξετάζω τον ρόλο των πολιτών και των καταναλωτών μέσα στην εσωτερική αγορά θεωρώ ότι οι Ευρωπαίοι καταναλωτές και πολίτες είναι η κεντρική αρτηρία για την λειτουργία μιας καλώς λειτουργούσας εσωτερικής αγοράς. Αυτό το έργο, να εμπλακούν οι πολίτες και οι καταναλωτές στην αναζωογόνηση αυτού του εγχειρήματος δεν θα είναι εύκολο. Μια και σε μεγάλο βαθμό οι κανονικοί πολίτες όσον αφορά την θεώρηση και γνώση της εσωτερικής αγοράς είναι σε χαμηλά επίπεδα ή ίσως και ανύπακτη η γνώση. Σαν αποτέλεσμα πρέπει να βρούμε τρόπους να αλλάξουμε την αντιμετώπιση των πολιτών και την οτροπία τους και να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη τους στην εσωτερική αγορά επειδή θα μπορεί να προστατεύει τα συμφέροντα και τις ανάγκες τους. Επίσης, η προστασία καταναλωτών στην έκθεσή μου θεωρώ ότι πρέπει να είναι προτεραιότητα στο, ε, στον ιστό της ε, νομοθετικής μας προσπάθειας ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διατύπωση αυτής της νομοθεσίας θα απαιτήσει από τους νομοθέτες να προσαρμοστούν σε ένα νέο υπόδειγμα, σε ένα νέο πρότυπο δράσης, ώστε να αποτελέσουν οι πολίτες μέρος του συστήματος ελέγχων, ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά η εσωτερική αγορά θεωρώ ότι μία από τις ε, κύριες ε, ανησυχίες μου και μελήματά μου είναι ότι κανένας ε, δεν ανέλαβε το εγχείρημα μέχρι τώρα να περιγράψει και να αναλύσει τα μη τεχνικά προσκόμματα και εμπόδια που αντιμετωπίζει η εσωτερική αγορά για την αναζωγόνηση της οικονομίας. Ένα από τα προβλήματα φαίνεται να είναι ότι η εσωτερική αγορά δεν προεκτείνεται και δεν δίνει την εικόνα ενός ολοκληρωμένου εγχειρήματο. Πράγματι, συζητάμε διαφορετικές οδηγίες, κανονισμούς και εκθέσεις. Υπάρχουν χιλιάδες τέτοια διαφορετικά νομοθετήματα και διατάξεις ε, που βρίσκονται διάσπατα σε διαφορετικές γενικές διευθύνσεις. Προσδοκώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναλάβει σοβαρή δράση ώστε να συντονιστεί το έργο, ώστε η στρατηγική 2020, η έκθεση Μόντι, η έκθεση Γκονθάλετ να συμπληρωθούν, να συντονιστούν και να ενταχθούν σε μια ενιαία στρατηγική για την επίτευξη τη ολοκλήρωση εσωτερική αγορά. Μεγάλα τμήματα τη ε, έκθεσή μου απορρέουν και αφορούν συγκεκριμένε προτάσει για την οικοδόμηση μια λειτουργούσα και αποτελεσματική εσωτερική αγορά. Για να επιβιώσει η εσωτερική αγορά πρέπει Ευρώπη να αναπτύξει στρατηγικές που θα δώσουν την ευκαιρία οι αγορέ να είναι οι καταλήτε για την οικονομική ανάκαμψη και ταυτόχρονα θα γίνει δεκτή αυτή η προσπάθεια από τους πολίτε και θα θεωρήσουν ότι προστατεύονται τα συμφέροντά τους και τα δικαιώματά τους. Η έκθεση προτείνει ένα σύνολο νομοθετικών και μη νομοθετικών προτάσεων για να αναζωογονήσουμε την ενιαία εσωτερική αγορά. Οι νομοθετικές προτάσεις συμπεριλαμβάνουν αρκετές ε, πολυάριθμες πτυχές όπως ε, τα τέσσερις, τις τέσσερις φάσεις ε, πρώτα απ' όλα την ενδιάμεση αναθεώρηση της ε, σημερινής κατάστασης δεύτερον την παγίωση και εδραίωση και συντονισμό όλων των διαφορετικών μέτρων, βελτίωση της εσωτερικής αγοράς και για μακροπρόθεσμη προοπτική είναι αναγκαίο να μην βασίσουμε όλες τις στρατηγικές μας στην ε, στρατηγική του 2020 και στην οικονομική κρίση και για να ζητήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει μια πρόταση για ένα νομοθετικό πακέτο μέτρων για την εσωτερική αγορά που θα συνδυάζει βραχυπρόθεσμα μέτρα με την μακροπρόθεσμη προοπτική και όραμα. Σε ένα άλλο επίπεδο, <clears throat> στις μη νομικές προτάσεις, όπως την Χάρτα των Πολιτών, που συμπεριλαμβάνει τις διαφορετικές προοπτικές να ζει κανείς οπουδήποτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μια στοχοθετημένη στρατηγική επικοινωνίας βασιζόμενη στις ανάγκες των πολιτών μας και άλλες τέτοιες δραστηριότητες θα διασφαλίσουν από κοινού ότι οι πολίτες θα αισθάνονται ότι εμπλέκονται και ότι δρούν όλοι από κοινού για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. Αυτή η νοοτροπία θα μας επιτρέψει πιστεύω να επεκταθούμε πέρα από τις παραδοσιακές ατραπούς και να μπορέσουμε περισσότερο να προσεγγίσουμε τους καταναλωτές, τους πολίτες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εκείνοι που θα κερδίσουν θα είναι εκείνοι που θα κατανοήσουν και θα αντιληφθούν το μεταβεβλημένο αυτό περιβάλλον και τις μεταβολές όσον αφορά τις δομές και τις τεχνικές προβλέποντας τις αλλαγές του μέλλοντος. Θέλω τέλος να τονίσω ότι η διαδικασία της ολοκλήρωσης της αγοράς δεν θα έπρεπε να θεωρείται δεδομένη ιδιαίτερα σε ένα από τα πιο ευαίσθητα χρονικά σημεία και πιο ευάλωτα χρονικά σημεία της ιστορίας για την εξέλιξη και ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. Στεναρά πιστεύω ότι η αναζωογόνηση και νέα καθέλκυση της εσωτερικής αγοράς πρέπει με συνεκτικό τρόπο και συντορισμένο τρόπο να ξεκινήσει. Θα πρέπει να συνδυάζεται όμως και με ευαισθησία, με πρακτικό πνεύμα. Και όπως είπε ο Jacques Delors, με ένα πνεύμα συνεργασίας και έκφρασης αλληλεγγύης αναμεταξύ μας. Γνωρίζω ότι υπάρχει ένας ε, αριθμός σημαντικών τομέων που θα έπρεπε να θεωρείται σημαντικό για την ολοκλήρωση τη εσωτερική αγορά. Όμω δεν μπόρεσα να καλύψω αυτόν τον τομέα πιο ε, εξειδικευμένα στην έκθεσή μου, γιατί είτε βρίσκεται αυτό ο τομέα εκτό αρμοδιοτήτων τη κοινοβουλευτική μα Επιτροπή ΙΝΚΟ ή πέρα από την εντολή που μου δόθηκε από την Επιτροπή μα ε, για να συντάξω αυτή την έκθεση, ή καλύπτονται αυτά τα σημεία από άλλε εκθέσει τη ΙΝΚΟ. Η έκθεση, όπω είπα πιο πριν, προτείνει να υιοθετήσουμε ένα νέο πρότυπο πολιτικής νοοτροπίας και προσέγγισης και θέλω να το τονίσω αυτό το σημείο με προστασία των καταναλωτών και την κοινωνική διάσταση που θα βρίσκονται στο επίκεντρο της διαδραμάτισης των ρόλων ε, σε αυτή την προσπάθεια. Όπω και είπα πιο πριν, δεν θεωρώ ότι είναι μια ε, αμετάκλητη διαδικασία και το ότι στο status quo στην εσωτερική αγορά θα πρέπει να αμφισβητηθεί και όλα να, ε, όλα να αποτελέσουν ε, ε, θέματα προβληματισμού και τίποτα να μην θεωρείται δεδομένο. Υπάρχουν εδώ αντιφάσεις, υπάρχουν ευάλωτα σημεία, υπάρχουν μεταβολές. Αυτές είναι πραγματικότητες. Πρέπει όμως αυτές τις πραγματικότητες να μπορέσουμε να τις μετατρέψουμε σε κίνητρα για να μπορέσει να υπάρξει ανάκαμψη και πρόοδος. Θέλω να ευχαριστήσω τους εισηγητές όλους για τις σημαντικές τις συνεισφορές για τη σύνταξη της έκθεσης καθώς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις προτάσεις της που θα προσπαθήσουμε να λάβουμε υπόψη. Θέλω τέλος να ευχαριστήσω τη γραμματεία, ιδιαίτερα Βάλτερ Τζοντάνα και τους συναδέφους για τις συνεισφορές τους. Ευχαριστώ. Well, Louis, thank you uh, very much Ευχαριστώ πολύ για την σαφέστατη παρουσίαση και για την έκθεση που είναι ιδιαίτερα πλούσια και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να αντλήσουμε από αυτό το πλούτο στις συζητήσεις μας. Και νομίζω ότι θα υπάρξει και καλή συνεισφορά και από τον κύριο Μόντι και από την Επιτροπή. Θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση τώρα, όμως θα σταματήσουμε στις 10 για την ψηφοφορία και όσοι έχουν απομείνει στον κατάλογο ομιλητών θα συνεχίσουν αργότερα μετά τις ε, ψηφοφορίες και μετά τον κύριο Μόντι. Ξεκινάμε με τον κύριο Σφάμπ, εκ μέρους του Σκιώδη Συγητή. Κύριε Σβάμπ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν, φυσικά θέλω εξ ονόματος της κοινοβουλευτικής μου ομάδας και εξ ονόματο του Γιώργου εισηγητού κυρίου Ατμακάρας που δυστυχώ δεν μπορεί να παραστεί να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την έκθεση. Είναι ένα πολύ καλό έγγραφο που σημαντικά στοιχεία δίνει για την ενιαία εσωτερική αγορά για τα επόμενα χρόνια. Και είναι μεγάλη χαρά για μα ότι είσαστε εσεί εδώ καθηγητά Μόντι. Έχουμε συναντηθεί και ο στόχο είναι να υπάρξει ένα New Deal, μια συμφωνία για την εσωτερική αγορά, να προταθεί μια νέα συμφωνία, ένα New Deal στους πολίτες και είναι ευτυχές το χρονικό αυτό σημείο της συνάντησής μας μαζί σας. Αν μου επιτρέπετε όμω, ίσω εξ ονόματο του συναδέλφου Κάρα, που όπω είπα δυστυχώ δεν μπορεί να παραστεί, καταρχήν δύο κύρια σημεία θα ήθελα να αναφέρω και μετά μια αξιολόγηση, προσωρινή αξιολόγηση να κάνω. Θα ήθελα να πω όμω πρώτα ότι για την, τροπολο... της ε, προθε... την ε, εκπνοή ε, της προθεσμίας για τροπολογίες στις 12 Απριλίου έλεγα ότι θα έπρεπε να παραταθεί ακόμα παραπέρα ώστε να υπάρξει δυνατότητα καθάθεσης τροπολογιών και να εμπλουτιστεί η έκθεση. Ιδιαίτερα αυτές οι τέσσερις φάσεις για την αναζωογόνηση της εσωτερικής αγοράς ενδιάμεση αναθεώρηση, παγίωση, βελτίωση και ανάπτυξη των μέσων και μακροπρόθεσμο όραμα για την εσωτερική αγορά είναι ένα ε, μια προσέγγιση που υπό το πρίσμα του ΕΛΚ για τη σημασία της εσωτερικής αγοράς στην Ευρώπη για τους καταναλωτές και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι σίγουρα ότι, σίγουρο ότι εξυπηρετεί και είναι καλό. Καθώς επίσης ε, και οι 20 πηγές για την εσωτερική αγορά που ε, την δυσαρέσκεια των πολιτών θα πρέπει να την αντιμετωπίσει είναι μια πρόταση που είναι πραγματικά πολύ θετική και με θετικό τρόπο γίνεται δεκτή. Ούτως ή άλλως όπως η αλλως οπω η προσέγγιση για την αντιμετώπιση τη εσωτερική αγοράς που τη συμμεριζόμαστε εμεί. Το θέμα του αν χρειαζόμαστε μια οδηγία πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών γενικού συμφέροντο είναι ένα θέμα που με μεγάλη προσοχή πρέπει να αντιμετωπιστεί. Διότι ένα πράγμα είναι σαφέ. Μπορεί, αν γίνει σωστά, να οδηγήσει σε μεγαλύτερη νομική ασφάλεια. Όμω ο κίνδυνο που είναι πάρα πολύ μεγάλο ελοχεύει και που τον αναγνωρίζουν τον κίνδυνο αυτό όλοι οι εμπλεκόμενοι ότι να υπάρξει μεγαλύτερη δηλαδή ενδεχόμενα γραφειοκρατία από ό,τι προτερήματα. Αυτό πρέπει να το αποφύγουμε. Γι' αυτό το, γι αυτό, αυτό το σημείο πρέπει να το βελτιώσουμε κάπω. Η εσωτερική αγορά, έτσι μου είπε και σημείωσε ο Μακάρας υφίσταται όχι μόνο από την ελευθερία των προσώπων που είναι όλο και πιο σημαντική και γι' αυτό σωστά θέτει το κέντρο βάρου η έκθεση σε αυτό το σημείο, αλλά επίση και στην ελευθερία διακίνηση των αγαθών, των εμπορευμάτων και χαιρόμαστε ιδιαίτερα ότι στην έκθεση εμπεριέχεται η πρόταση μια πιο αυστηρή, ένα πιο αυστηρό, πιο αποτελεσματικό και γοργό έλεγχο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να γίνεται για την ε, εφαρμογή από τα κράτη-μέλη ε, τη οδηγία και των διατάξεων για την ελευθερία διακίνηση των αγαθών αυτή η πιο αυστηρή ας το πω έτσι προσέγγιση κατά πόσον μπορεί με μια πιο φιλική δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συνδυαστεί που όπως είπε ο καθηγητής Μόντι αφορά τα social welfare ε, δηλαδή τα θέματα της, ε, του κράτους της κοινωνικής ευημερίας και τα προτερήματα της ευημερίας κατά πόσον δηλαδή θα μπορέσουμε να τα εκμεταλλευτούμε αυτά και θα πρέπει εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δραστηριοποιηθεί για να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες παρόλα αυτά πιστεύω ότι η πιο γοργή, πιο αποτελεσματική ε, διαμόρφωση διαμόρφωση των διεργασιών και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο πρέπει να διασφαλιστεί ώστε η υλοποίηση των υφιστάμενων δικαιωμάτων στο τέλος τέλος να μπορέσει να λειτουργήσει με το σωστό τρόπο. Το θέμα τώρα του οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες πρέπει ή όχι να ενταχθούν στην ε, έκθεση. Εσείς είπατε ότι κύριε Γκρέκ ότι υπάρχει και έργο άλλων κοινοβουλευτικών επιτροπών που εμπλέκονται εδώ. Το θέμα είναι αν μπορούμε να πούμε κάτι για τον εναρμονισμό φορολογικών θεμάτων ως ευκαιρία για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. Το θέμα είναι αν η έρευνα και η καινοτομία θα έπρεπε να τονιστεί ιδιαίτερα. Γνωρίζουμε ότι βρισκόμαστε σε παγκόσμιο ανταγωνισμό και αυτό το είπατε κι εσείς με σαφήνεια. Στόχος της ε, ενιαίας εσωτερική αγοράς πρέπει να είναι στο διεθνή ανταγωνισμό η Ευρώπη μακροπρόθεσμα να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο. Η οικονομική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια ήταν πλην, ε, συν 8% στην Κίνα, μείον 5% στην Ευρώπη. Ακριβώς όμως ως εκπρόσωποι της νέας γενεάς πρέπει να πούμε ότι αυτό δεν είναι η σωστή προοπτική για το μέλλον. Πρέπει να επανέλθουμε να έχουμε τουλάχιστον εξίσου σημαντική ανάπτυξη οικονομική όπως της ΗΠΑ και αυτό να είναι κάτι το οποίο θα διαμορφώσει θετικά την, ε, των δύο των Ευρωπαίων πολιτών. Δεν θέλω να αναφερθώ σε όλα τα σημεία. Στι συλλογικέ προσφυγέ εδώ ε, επιθυμεί ο εισηγητή μια ισορροπημένη προσέγγιση. Ε, θέλει οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αναφέρονται σωστά. Βλέπω ότι σε πολλά σημεία έχει γίνει αυτό. Ολοκληρωμένα πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή βάση εργασίας αυτή. Και έτσι έτσι μπορούμε να καθορίσουμε τη θέση μας ε, στην ε, Επιτροπή μας ε, για την εσωτερική αγορά. Ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ άλλη μια φορά. Uh, uh, Ευχαριστώ κύριε Σφάπ. Κύριε Ρόσφολ. Ευχαριστούμε τον Λουί Γκρέφ για την εξαιρετική έκθεση και για τις τον τρόπο με τον οποίο ακούσατε και τους σκιώδεις συζητητές και όλους τους ευρωβουλευτές. Επίσης θα ήθελα να συγχαρώ τον ε, κύριο Χάρμπορ για την συνάντηση που διοργανώσατε σήμερα και με τον καθηγητή τον κύριο Μόντι. Εδώ θα ήθελα να επανέλθω στα πρακτικά του Στρασβούργου στις 14 Δεκεμβρίου πέρυσι που πάλι είχε έρθει ο κύριος Μόντι και βλέπω ότι υπάρχει σύγκληση σε αυτά που λέγατε όσον αφορά την συνολική, την ολιστική προσέγγιση που χρειάζεται. Είναι ένας τρόπος να πούμε ότι η ενιαία αγορά δεν αποτελείται από πολλά μικρά αλλά από ένα συνολικό όραμα που θα σημαίνει φορολογική και βιομηχανική πολιτική, κοινωνική πολιτική και πολιτική προστασία των καταναλωτών μεταξύ άλλων, όπως αναφέρει και ο κύριος Γκρέ στην έκθεσή του, όπου αναφέρεστε στο σεβασμό των πολιτών, κυρίως των πολιτών και μετά των καταναλωτών. Επίσης ε, πρέπει να συμπεριληφθεί και ο περιβαλλοντικός ε, παράγοντας ε, αλλά και τα κοινωνικά θέματα, ειδικά υγεία. Και εδώ θα ήθελα να επισημάνω κάποια πράγματα επί της ουσίας. Όπως μας είπατε ότι δεν υπάρχει πλέον εμπιστοσύνη όσον αφορά την ενιαία αγορά. Εντάξει υπάρχει η κρίση αλλά αυτό προϋπήρχε της κρίσης Γνωρίζουμε επίσης ότι η οδηγία για τις υπηρεσίες δεν βοήθησε την ε, αλληλοκατανόηση πολιτών και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει και εκεί λοιπόν να πούμε τα ίδια πράγματα, ειδικά όσον αφορά τα κοινωνικά θέματα και τα θέματα υγείας. Θεωρώ ότι η υγεία δεν είναι ένας οικονομικός τομέας όπως οι υπόλοιποι και δεν μπορούμε να την ενσωματώσουμε έτσι απλά στην ενιαία αγορά παρόλο που υπάρχουν πράγματα που μπορούν να βελτιωθούν ειδικά όσον αφορά την διασυνοριακή κατανάλωση περίθαλψης υγειονομικής. Και κάτι όσον αφορά τον ορισμό της ε, ενιαίας αγοράς. Χρησιμοποιούμε τον κλασικό ορισμό των οικονομολόγων που έχει να κάνει με ποσότητες και τιμές. Έχουμε δηλαδή έναν αυστηρό ορισμό της ενιαίας αγοράς. Τότε θα ήταν επικίνδυνο να διευρύνουμε την ενιαία αγορά στο κοινωνικό τομέα και το τομέα της υγείας. Ή έχουμε μια πιο ευρία έννοια για το τι σημαίνει ενιαία αγορά που έχει να κάνει με την ε, κοινωνική οικονομία της αγοράς και εκεί περνάμε πέρα από έναν ορισμό που, των οικονομολόγων και μπορούμε άρα να συμπληρώσουμε θέματα όπως η υγεία και ο, και ο κοινωνικός τομέας. Πρέπει να το δούμε αυτό το θέμα και το, να το εξετάσουμε. Και είναι πιθανόν ότι η απάντηση δεν θα είναι ούτε αποκλειστικά η μία ούτε αποκλειστικά η άλλη. Σε κάθε περίπτωση πάντως πρέπει να προσέξουμε ώστε να μην χάσουμε τη δημοκρατία και να μην βλεχτούμε στη γραφειοκρατία. Το δεύτερο θέμα. Θέλουμε να ξαναδώσουμε ελπίδα στους σε όλους τους μετόχους της εσωτερικής αγοράς εδώ. Όμως για να γίνει αυτό θα πρέπει να κάνουμε πολλά συγκεκριμένα θέματα και ίσως πρέπει να προσθέσουμε και άλλα. Για παράδειγμα, καταρχάς όσον αφορά τις επιχειρήσεις, ειδικά τις μικρομεσαίες, πρέπει να επανεξετάσουμε το θέμα της διανοητικής ιδιοκτησίας. Πρέπει να επανεξετάσουμε το θέμα των ευρωπαϊκών ευρεσιτεχνιών που θα μπορούσε να βοηθήσει πολύ την ανάκαμψη των επιχειρήσεων. Και υπάρχουν και πολλά που μπορούμε να πούμε και για το δημόσιο τομέα. Είχαμε και χτες μια πολύ ευαίσθητη συζήτηση για τις καθυστερημένες πληρωμές. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με την έννοια αγορά. Και κάτι ακόμη, όπως είπε και ο κύριος Σβάμπ προηγουμένως. Ναι, κύριε Γκρέσ, η δυσλειτουργία της ε, ενιαίας ε, αγοράς είναι ένα από τα 20 πρώτα θέματα που δημιουργούν έλλειψη ικανοποίηση στους πολίτες. Όμως, τι μπορούμε να κάνουμε για, να... για την αναγέννηση της ενιαίας αγοράς. Δεν χρειάζεται μόνο ενσωματωμένη οικονομία και η αντιμετώπιση του προστατευτισμού αλλά και θέματα όπως για παράδειγμα η αντιμετώπιση των κρατών που καθυστερούν στην εφαρμογή της οδηγίας. Και τέλος, ίσως πρέπει να δούμε το θέμα και από άποψη προοπτικής. Έχουμε προβλήματα δημογραφικά και γύρανσης και εδώ θα πρέπει να βοηθήσει η ενιαία αγορά. Πέρα από το περιβαλλοντικό θέμα πρέπει να δούμε τι θα μπορέσουμε να δώσουμε στον ευρωπαϊκό πληθυσμό υπό το βάρος του δημογραφικού προβλήματος. Επίσης, είπαμε ότι πρέπει να υπάρξει στοχευμένη διάδοση, όχι απλά προπαγάνδα υπέρ της οδηγίας. Πώς θα το κάνουμε αυτό. Ίσως να χρησιμοποιήσουμε διαφορετικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ενδεχομένως τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης αντί για τα μεγάλα μέσα. Και θα έπρεπε να εξετάσουμε ακριβώς τι μπορούμε να προσφέρουμε στον καταναλωτή και να δείξουμε στον καταναλωτή τι μπορούμε να κάνουμε. Να του στείλουμε πολύ συγκεκριμένα μηνύματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Πολύ καλά σημεία. Η κυρία Ρούλε στη συνέχεια, γιατί δεν είναι εδώ ο σκιώδης συζητητής σας και μετά μπορούμε να περάσουμε στον κύριο Γκυγιόν και μετά θα περάσουμε στις ψηφοφορίες. Κυρία Ρούλε παρακαλώ. Uh, Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την έκθεσή του και την καλή συνεργασία με όλες τις κοινοβουλευτικές ομάδες. Και νομίζω θέτει τα σωστά θέματα στο επίκεντρο. Θέλω να τονίσω για άλλη μια φορά πόσο το χαιρετίζω ότι οι καταναλωτές πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της ε, εσωτερικής αγοράς και του δίνω απόλυτο δίκιο. Αν θέλουμε να αποκαταστήσουμε το θέμα της σχέσης εμπιστοσύνης από τους καταναλωτές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να υπάρξει νομική βεβαιότητα και νομική ασφάλεια διαφορετικά δεν θα έχουμε τις ευθές επιπτώσεις. Το βρίσκω σημαντικό το θέμα των χρηματοοικονομικών αγορών για άλλη μια φορά να καλυφθεί, να ε, θυγεί εδώ, διότι είναι απόλυτα αναγκαίο για την εμπιστοσύνη των πολιτών που ακόμα δεν είναι δεδομένη και πρέπει εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση να υποβάλει προτάσεις και να δράσει. Τι θα γίνει σε σχέση με την ε, απελευθέρωση των ε, χρηματοοικονομικών αγορών, να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη, να διασφαλιστούν τα μελήματα των καταναλωτών και έτσι προστατευτούν οι καταναλωτέ. Θέλω να υπενθυμίσω ότι πριν από αυτή την κρίση των χρηματοοικονομικών αγορών είχαμε προβλήματα στον οικονομικό τομέα και υπήρχαν σκάνδαλα, διότι υπήρχε μειωμένη προστασία καταναλωτών. Κάτι πρέπει να γίνει λοιπόν. Ω πράσινη θέλω να πω ότι το θέμα τη ενέργεια, των κλιματικών αλλαγών δεν, δεν καλύπτεται πλήρω. Κάτι παραπάνω πρέπει να κάνουμε, ώστε μέχρι το τέλο ε, τη προθεσμία για κατάθεση τροπολογιών να καταθέσουμε κάποιε τροπολογίε να συμπληρωθεί αυτό ε, ο τομέα. Διότι η μεγάλη πρόκληση είναι το θέμα των κλιματικών αλλαγών και το θέμα πώς μπορούμε να συνεισφέρουμε σε καλύτερη απόδοση και εκμετάλλευση των ενεργειακών πόρων. Εγώ πιστεύω ότι αυτά είναι κέρια ε, θέματα για τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν σωστά όσον αφορά το μέλλον μας και πρέπει να αναφερθούν αυτά πιστεύω. Ένα επιπλέον σημείο που θα ήθελα και πιστεύω ότι ε, θα ήθελα να πω ότι δεν καλύπτεται επαρκώς είναι ο τομέας ε, των παροχών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος. γίνεται αναφορά αφορά στην ε, οδηγία πλαίσιο. Όμω το θέμα έχει μεγαλύτερη εμβέλεια. Το θέμα είναι η εμπιστοσύνη στην εσωτερική αγορά. Αν η εσωτερική αγορά έχει πολύ μεγάλο βάθο ε, παρέμβαση στι τοπικέ οικονομίε, ε, αν υπάρχει αυτό το βάθο στι παρεμβάσει στι κοινωνικέ υπηρεσίε, τότε σε πολλού πολίτε θα δημιουργηθεί απώλεια εμπιστοσύνη και θα δημιουργηθεί αβεβαιότητα. Η Ευρώπη έχει ένα πρότυπο μεικτή οικονομία. Από τη μία πλευρά έχουμε οι μεγάλε ισχυρέ ε, ιδιωτικέ επιχειρήσει. Από την άλλη πλευρά όμω έχουμε ικανοποιητικέ προσφορέ υπηρεσιών από τον δημόσιο τομέα στι υπηρεσίε. Εδώ πολλά έχουν διολυστήσει τα τελευταία χρόνια και έχουν ε, α το πω έτσι αποσυναρμολογηθεί. Είναι σημαντικό, δεν ξέρω το τι θα γίνει με την ε, οδηγία πλαίσιο, πρέπει να μειωθεί η πίεση όσον αφορά τι υπηρεσίε καθολικού συμφέροντος. Κάτι πρέπει να γίνει και σε αυτόν τον τομέα. Και τώρα για το θέμα των δικαιωμάτων δικαιωμάτων ε, όσον αφορά την ε, παροχή υπηρεσιών, το βάθος παρέμβασης ε, οδηγεί σε μεγάλη γραφειοκρατία, σε μεγάλη αβεβαιότητα των πολιτών. Πρέπει να εξεύρουμε μια σωστή ισορροπία, αφενός μεταξύ επικουρικότητας και από την άλλη πλευρά μεταξύ εσωτερικής αγοράς. Uh, um, Ευχαριστώ κύριε Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε όπως και οι υπόλοιποι, θα ήθελα και εγώ να πω ότι ήταν θαυμαστό το έργο του Λουί Γκρέγκ γιατί ήταν δύσκολο το θέμα και περιέλαβε πολλές διαφορετικές συστάσεις σε λίγες σελίδες. Αλλά επίσης και γιατί είχαμε πολύ καλή ατμόσφαιρα συνεργασίας με τον κύριο Γκρέχ, όλοι οι σκιώδεις εισηγητές. Συμφωνώ με τους βασικούς άξονες του κυρίου Γκρέχ. Πρώτος άξονας πρέπει να είναι η ισότιμη μεταχείριση στην εσωτερική αγορά, το level playing field. Είναι σημαντικό αυτό, δηλαδή οτιδήποτε επί του οποίου συμφωνούμε πρέπει να εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, υπάρχουν κάποια θέματα όπως ε, η διανοητική ιδιοκτησία, η περιφερειακή ανάπτυξη, το περιβάλλον ε, και τα λοιπά που θα μπορούσαν να τονιστούν περισσότερο, χωρίς να θέλω να επικρίνω την έκθεση. Και περνάω στο θέμα που ενδιαφέρει ιδιαίτερα την ομάδα μου πώς θα μπορέσουμε να αγγίξουμε τις καρδιές και την ψυχή των ανθρώπων. Δεν νομίζω ότι μια ανακοίνωση από τις Βρυξέλλες είναι η απάντηση. Γνωρίζω ότι στη χώρα μου οι άνθρωποι δεν εντυπωσιάζονται ιδιαίτερα όταν βλέπουν καινούριους φακέλους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουν να βλέπουν αποτελέσματα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα πολύ πρακτικό. Αυτή τη στιγμή ακούω πολλά παράπονα από ανθρώπους που θέλουν να πάνε στην Γερμανία και να ψωνίσουν, αλλά όταν πάνε σε ένα ATM τράπεζας πρέπει να πληρώσουν 5 ευρώ για να κάνουν ανάληψη. Εκεί υπάρχει κάποιο πρόβλημα και πρέπει να το εξετάσουμε σε συνεργασία και με τις οργανώσεις καταναλωτών. Αυτό δεν είναι παρά ένα παράδειγμα. Όμως αυτό το παράδειγμα χαλάει τόσα πολλά στην πράξη που όποια ανακοίνωση και όποια στρατηγική να κάνουν οι Βρυξέλλες δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό το βασικό πρόβλημα που έχουν οι άνθρωποι στα ψώνια τους στο εξωτερικό. Τώρα, όσον αφορά τους κανόνες που ισχύουν αυτή τη στιγμή για τους εργαζόμενους, τους μισθωτούς, Υπάρχουν πολλά προβλήματα αυτή τη στιγμή. Διαπιστώνω ότι όταν έχουμε εργαζόμενους από άλλα κράτη-μέλη δεν εργάζονται υπό τις ίδιες συνθήκες γιατί δεν είναι αρκετά αποτελεσματική η έλεγχη επιθεωρήσεις και επίσης γιατί στα κράτη-μέλη μας δεν έχουν αναπτυχθεί ακόμη τόσο οι διαδικασίες για τις επιθεωρήσεις. Αν όμως δεν υπάρξει σεβασμός αυτών των κανονισμών δεν θα έχουμε πραγματική ελευθερία μετακίνησης. Κάτι άλλο τώρα. Ε, υπάρχουν πολλά παράπονα για τις Βρυξέλλες και υπάρχουν και εθνικές έρευνες δείχνουν ότι όταν εναρμονίζουμε κάτι, ορισμένες φορές δημιουργούμε κανόνες που δεν είναι ιδιαίτερα θετικοί για τις επιχειρήσεις που θέλουν να δραστηριοποιούνται μόνο τοπικά. Πρέπει λοιπόν να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ του πώς μπορούμε να βοηθήσουμε την ιανιαία αγορά και πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη γραφειοκρατία που προκύπτει. Πάντως πρέπει να υπάρχει συνοχή στην εσωτερική αγορά για τους πολίτες, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επίσης για τους εργαζόμενους. Και νομίζω ότι αυτά μπορείτε να τα συμπεριλάβετε κύριε Γκρέχ με τη βοήθεια και του κυρίου Μόντι. Λοιπόν, ε, ευχαριστώ ε, κύριε Διό. Ε, επειδή εγώ είμαι ο μόνος που δεν παρενέβη. Θα ήθελα να κάνετε λίγο υπομονή και να παρουσιάσω ορισμένα σχόλια πριν προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Θέλω να ευχαριστήσω τον Λουί Γκρέκ, ιδίω διότι, ε, διότι είχε εκτενήσει συζητήσεις με όλους τους χειώδεις εισηγητές προηγουμένως και χαιρόμαστε γιατί οι ιδέες έχουν περιληφθεί στην έκθεση και αυτό είναι θετικό. Από πρακτικής απόψεως, έχοντας δει τις αντιδράσεις, επίσης Πιστεύω ότι θα έπρεπε να συζητήσουμε το Λουί τη δυνατότητα να έχουν περισσότερο χρόνο για τροπολογίες οι συνάδελφοι διότι υπάρχουν τόσα θέματα ώστε θα χρειαστείτε ίσως περισσότερο χρόνο και θα εκτιμήσετε την επέκταση της προθεσμίας και θα μπορέσει και ο Λουί να σεβαστεί τις προθεσμίες που έχει θέσει στον εαυτό του. Άρα ε, αυτό μπορεί να συζητηθεί είτε πριν είτε μετά τη τις ψηφοφορίες. Υπάρχουν ορισμένες βασικές συστάσεις. Ε, σε μια τέτοια έκθεση σαν του Λουί Γκρέκ όπου έχει ε, απαριθμίσει τι είναι εφικτό είναι το θέμα ε, που θα πρέπει να μας απασχολήσει για να μπορέσουμε να έχουμε αποτελεσματικές προτάσεις και πολύ χαίρομαι διότι έχει συγκεντρώσει όλες τις πτυχές της εργασίας την οποία κάνουμε κάνουμε εδώ και θέτει τους καταναλωτές και τους πολίτες στο επίκεντρο του τι πρέπει να προσφέρει η ενιαία αγορά. Και ορισμένες από τις ε, καθημερινές ενοχλήσεις ε, των πολιτών ε, σε τομείς όπως τα τέλη που πληρώνουν για τα μηχανήματα από τα οποία παίρνουν χρήματα μαυρίζουν την εικόνα της ενιαίας αγοράς γιατί αυτό που μας λένε από το ε, επεξεργάζεστε αυτό το πρόγραμμα και δεν μπορείτε να μας δώσετε αυτό το οποίο θα έπρεπε. Δηλαδή ε, απλά πράγματα τα οποία δεν είναι δύσκολα. Οπότε η ιδέα του Λουίς ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, ε, κάνει αυτή την ε, άσκηση, να καθορίσει δηλαδή τις, τα 20 πιο εκνευριστικά στοιχεία για τους πολίτες στην ενιαία αγορά, θα μας δείξει ότι ακούμε τις ανησυχίες των πολιτών σχετικά με την ενιαία αγορά. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι ένα θέμα το οποίο ε, πρέπει να περιληφθεί στη στρατηγική της Επιτροπής και ο Επίτροπος Μπανιέ την εποχή που ήταν μέλος αυτής της Επιτροπής είχε διαπιστώσει ότι η ενιαία αγορά δεν πρέπει απλώς να θεωρείται σαν γραφειοκρατική εφαρμογή των κανονισμών αλλά ουσιαστικά πρέπει να προασπίζεται ε, το, ε, τους πολίτες ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όπως είπε και η κυρία Ρούλε υπάρχουν βασικά θέματα για την ε, περιβαλλοντολογική, επιτροπή, ε, ε, περιβαλλοντολογική πολιτική για την χρήση των, των πόρων βασικά πράγματα και νομίζω ότι η κυρία Ρέντινγκ είναι ο σύμμαχός μας σε αυτά τον περασμένο μήνα όταν είχε έρθει σε αυτή την Επιτροπή ε, είχε εκφραστεί πολύ θετικά και μαζί με τον κύριο Μπανιέ έχουμε τώρα δύο συμμάχους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, θα χρειαστεί λοιπόν ένα είδος μανιφέστο για την ε, ενιαία αγορά το οποίο θα απευθύνεται στους πολίτες. Για να ενισχύσουμε τη θέση μας λοιπόν όταν συζητάμε με τα Εθνικά Κοινοβούλια και τα κράτη-μέλη σχετικά με την ενιαία αγορά θα πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτές τις λύσεις διότι έχουν γίνει ακροάσεις για μελλοντική νομοθεσία προβλέπουμε ακρόαση για την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας όπως η οδηγία για την παροχή υπηρεσιών και θα πρέπει να ενθαρρύνουμε και τους άλλους συναδέλφους να πάρουν σοβαρά τα θέματα αυτά αλλά επίσης υπάρχουν προσπάθειες που πρέπει να καταβληθούν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και εχθές ε, συζητούσαμε τον πρόεδρο του Συμβουλίου για τα αποτελέσματα της διασκέψεως κορυφής γιατί τα αποτελέσματα και τα πορίσματα αυτού του Συμβουλίου ήταν απογοητευτικά σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισαν τα θέματα ενιαίας αγοράς και όχι μόνο και εκπαίδευσης και επίλυσης των θεμάτων φτώχειας που είναι πολύ σημαντικά και θέματα πρέπει να υλοποιηθούν αλλά η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς και η επίλυση των προβλημάτων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των καταναλωτών δεν αναφέρεται καν στα συμπεράσματα και ε, υποθέτω ότι δεν συζητήθηκαν καθόλου στο Συμβούλιο. Είναι λοιπόν ε, η ναυαρχίδα μας η οποία πρέπει ε, να προβληθεί για να μπορέσουμε να έχουμε πραγματικά πραγματικά ωφέλη για τους πολίτες, για τους καταναλωτές, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τις μεγάλες επιχειρήσεις στα πλαίσια της ενιαίας αγοράς για να υπάρξει μεταφορά ε, γνώσης η οποία είναι επίσης πολύ σημαντική. Αυτές είναι πρωτοβουλίες τις οποίες πραγματεύονται, ε, θα έπρεπε να πραγματεύονται οι εθνικές κυβερνήσεις οι οποίες όμως τώρα ασχολούνται με άλλα πράγματα. Δεν ε, προσπαθούμε να εφεύρουμε την ε, πυρίτιδα αλλά θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη αξία στα πράγματα που κάνουν οι πολίτες. Μπορούμε να βοηθήσουμε, μπορούμε να εφαρμόσουμε ορισμένα πράγματα με ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αντί να καταρτίζουμε ανέφικτους στόχους. Μπορούμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε προς το στόχο αυτή, αυτή την προσπάθεια και ίσως θα μας βοηθήσει και η έκθεση του Μάριο Μόντι οπότε θα έχουμε με μία διπλή γραμμή επιθέσεως για την επίλυση αυτών των θεμάτων. Υπάρχουν λοιπόν διάφορες προτάσεις οι οποίες είναι στον αέρα για το πώς μπορούν αυτά τα θέματα να εφαρμοστούν και ο κύριος Μόντι προτείνει και ένα νομοθετικό πακέτο. Μου αρέσει η φιλοδοξία του εδώ αλλά ε, δεν νομίζω ότι ουσιαστικά αυτό που χρειαζόμαστε είναι νέα νομοθεσία. Θέλω να κάνω στο Λουί μία πρόταση τώρα στον εισηγητή, διότι έχουμε ένα προηγούμενο όπου έχουν δεχτεί το Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη ότι δηλαδή ε, ε, εάν υπάρξει, εάν υπάρξει ένα συνδυασμός πρωτοβουλειών με ισχύουσα νομοθεσία να έχουμε μία πράξη a single market act μία πράξη ενιαίας αγοράς και ουσιαστικά αυτό πρέπει να ζητήσουμε ένα τέτοιο έγγραφο το οποίο θα συνδυάζει και τις ιδέες για νομοθεσία αλλά και τις μη νομοθετικές πρωτοβουλίες πρωτοβουλίες και που θα βοηθήσει τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να εφαρμόσουν την νομοθεσία που είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί και μας ενοχλεί. Και όπως είπε πολύ σωστά ο Λί θα πρέπει να ε, διαθέσουμε περισσότερες πληροφορίες. Όπως είπε ο κύριος Ροσφόρ, υπάρχουν πολλές ιδέες που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, με μελέτε περιπτώσεων, ένα blog ενίας αγοράς όπου ο καθένας θα μπορούσε να καταγράφει τις ανησυχίες του και τα θέματα που τον ενοχλούν, διότι ε, ακόμη και στο iPhone μπορεί κανείς να περάσει τα 20 βασικά θέματα της ενιαίας αγοράς. Και αν δείτε ε, ε, τα παράπονα που έρχονται σχετικά π.χ. με το Solvit ε, και την κλίμακα του προβλήματος αυτού διαπιστώνουμε ότι είναι τεράστια, δεν το επιλύουμε και η οδηγία για την παροχή υπηρεσιών και η αμοιβαία αξιολόγηση είναι μια ιδέα που μας λέγει ότι υπάρχουν και άλλοι τομείς όπου θα πρέπει να εφαρμοστεί η νομοθεσία νέας αγοράς. Διότι το πρόβλημα που τίθεται είναι ότι αναπτύσσουμε νέες ιδέες σε διάφορα σε διάφορους χώρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χωρίς όμως να συνδυάζουμε ε, μεταξύ των προσπαθειών τις κινήσεις οι οποίες γίνονται. Θα έπρεπε λοιπόν ε, ίσως να αποστασιοποιηθούμε και να πούμε ε, εάν έχουμε μία πηγή καλών ιδεών στο Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε επιχειρήσεις, στις κυβερνήσεις, στους πολίτες

Ας ε, ε, αναλάβουμε μία πολιτική πρωτοβουλία να χρησιμοποιήσουμε τα θέματα αυτά σε όλους τους τομείς για να έχουμε μία κοινή προσέγγιση, να επιλύσουμε τις, ε, τα παράπονα των πολιτών και των επιχειρήσεων που δεν θα έπρεπε πλέον να υπάρχουν μετά από τόσο καιρό και να μην υποθάλπουμε την πολιτική εικόνα του πώς προχωράμε. Νομίζω ότι αυτό είναι ο στόχος της έκθεσης αυτής και ε, ε, ο συνδυασμός με το τι κάνει ο Μάριο Μόντι θα μας βοηθήσει. Από τη μια πλευρά λοιπόν θα πρέπει να δώσουμε στους συναδέλφους χρόνο να συμβάλλουν αλλά από την άλλη πλευρά θα ήθελα να ψηφίσουμε ε, την έκθεση αυτή πριν από τη διάσκεψη κορυφή του καλοκαιριού πριν την παρουσίαση της εκθέσεως του Μάριο Μόντι γιατί πιστεύω πιστεύω ότι με αυτή τη βάση θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε πολύ καλά και ευχαριστώ τον Λουί Γκρέχ, τον εισηγητή, για τις προσπάθειές του. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Τώρα λοιπόν ξαβάζω το καπέλο μου του Προέδρου και ε, ε, αντί να συζητάμε για την εσωτερική αγορά ε, θα προχωρήσουμε στις δύο, στις δύο ψηφοφορίες για την ονομασία των κλωστοϊφαντουργικών και την διακυβέρνηση του διαδικτύου και ο Μάριο Μόντι θα πάει να πιει καφέ. Ελπίζω θα έχουμε τελειώσει ως τις 11 ε, ε, ό,τι και να γίνει θα σε περιμένουμε για τις 11 και νομίζω ότι αυτό θα είναι καλό. Έχετε όλοι τις κάρτες σας ψηφοφορίας. Για να προχωρήσουμε λοιπόν. Νομίζω ότι έχετε τις κάρτες σας τις οποίες θα χρησιμοποιήσουμε όταν είναι αμφίβολη η έκβαση της ψηφοφορίας. Ας κάνουμε λοιπόν έναν έλεγχο για να δούμε ποιος παρίσταται και ποιος ψήφισε. Λοιπόν, θέλω τώρα να παρακαλέσω όλα τα μέλη του ΕΛΚ οι οποίοι θα ψηφίσουν να ψηφίσουν τώρα για να ελέγξουμε ότι λειτουργούμε σωστά. Ελέγχουμε την ηλεκτρονική ψηφοφορία για τους ευρωβουλευτές του ΕΛΚ. Έχουμε 13 μέχρι στιγμής 14 14 Λοιπόν, 14 από το ΕΛΚ. Ε, οι σοσιαλιστές τώρα ψηφίζουν οι σοσιαλιστές ευρωβουλευτές έχουμε 12 ή 10 έπρεπε να έχουμε 10 και έχουμε 12 και 13 μάλιστα τώρα μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι θα ψηφίσουν μόνο 10 από τους σοσιαλιστές. Μετά έχουμε τους φιλελεύθερους. Παρακαλώ να ψηφίσουν οι φιλελεύθεροι. Ξεκινάει η ψηφοφορία για τους φιλελεύθερους. Τρεις, μπορείτε να, να έχετε και τέσσερις. Πράσινοι. τρει νομίζω. Ε, τρεις ε, Ευρωπαίους συντηρητικούς εκ των οποίων εγώ είμαι ένας. Οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε απλώς ε, ε, οι σοσιαλιστές να διασφαλίσουν ότι είναι εδώ οι 10 και θα δώσω τον λόγο στον εισηγητή ε, για το θέμα της ενιαίας αγοράς για τους καταναλωτές και τους πολίτες, τον κύριο Μάντερς. Μάλλον με συγχωρείτε, για την ονομασία των κλωστοεφαντουργικών, τον κύριο Μάντερς. Είχαμε πολλές ε, συμβιβαστικές τροπολογίες και μία μόνο βελτίωση. Προσπαθήσαμε να βελτιώσουμε την εσωτερική αγορά όπως θα ήθελε και ο κύριος Μόντι και συνδυάσαμε αυτή την οδηγία με την ε, πρόταση της οδηγίας του 2005 για τους τελωνιακούς κώδικες που μπλοκαρίστηκε στο Συμβούλιο και τη συνδυάσαμε και με τα παράγωγα ζωικών προϊόντων που συνδυάζεται με την οδηγία του 1994 για τα παπούτσια και ε, πρέπει να ε, δούμε ε, εάν ένα παπούτσι περιέχει δέρμα ή είναι όλο δερμάτινο και ο πολίτης και καταναλωτής δικαιούται να το γνωρίζει. Κατά τα άλλα ζητήσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει ορισμένες αξιολογήσεις επιπτώσεων σε ορισμένα θέματα ε, παραδείγματος, ε, χάρη παραδείγματος. Όχι δηλαδή ε, αποκλειστικά τα θέματα αυτά. Ίσως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωρίζει και περισσότερα θέματα και τους δίδουμε το πράσινο φως να εξετάσουν όλα τα θέματα και ενδιαφερόμενοι θα μπορέσουν να διατυπώσουν απόψεις, να τις στείλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν το κρίνει σκόπιμο θα διατυπώσει προτάσεις. Έχω μία τροπολογία για τον κύριο Κάρας. Εάν πάτε στον ράφτη για να φτιάξετε ένα κουστούμι, να ράψετε ένα κουστούμι, τότε αυτή η διεργασία αποκλείεται. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρξει μία προφορική τροπολογία γιατί ο κύριος Κάρας δεν είναι εδώ αλλά εγώ την έχω αναλάβει και κατά τα άλλα θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για ε, το ενδιαφέρον ταξίδι στο Μιλάνο και όλες ε, οι συμβιβαστικές προτάσεις έχουν ε, διεκπαιρεωθεί και η ομάδα σας κύριε Πρόεδρε ήταν πολύ συνέβαλε πολύ θετικά και ελπίζω θα συνεχίσουμε έτσι. Ένα τελευταίο όμως θέμα είναι η τελευταία τροπολογία η οποία αναφέρεται εις ε, τις διαπραγματεύσεις μετά από το νέο κώδικα συμπεριφοράς όπου πρέπει να ψηφίσουμε δηλαδή ότι έχουμε εντολή διαπραγματεύσεως με την Επιτροπή και το Συμβούλιο για να δούμε αν θα συμφωνήσουμε σε πρώτη ανάγνωση αλλά μπορεί να υπάρξει αυτή η ψηφοφορία από ό,τι κατάλαβα εχθές εις ε, τους συντονιστές και ελπίζω ότι θα υπερψηφίσετε την έκθεση αυτή για την εσωτερική ε, αγορά. Ευχαριστώ ε, και χαίρομαι ε, ότι ο ράφτης του κυρίου Κάρας θα εξαιρεθεί με την προφορική του τροπολογία δεν θα προτείνω να ψηφίσουμε ε, το διαδικαστικό γιατί δεν έχει συζητηθεί ε, με τους συντονιστές το θέμα αυτό αλλά πρώτα θα έπρεπε να συζητήσετε με το Συμβούλιο να δούμε κατά πόσον οι θέσει μας είναι, είναι ευθυγραμμισμένες και όπως είπε η κυρία Γκέφχαρτ ε, πολύ σωστά και συμφωνούμε όλοι οι συντονιστές αυτή της ε, ε, Επιτροπής θεωρούν ότι οι συμφωνίες πρώτης ανάγνωσης αποτελούν εξαίρεση και επειδή το θέμα αυτό κυκλοφορεί εδώ και κάμποσο καιρό δεν είναι κατάλληλο. Εάν όμως μας πείσετε ότι υπάρχει πλήρης ευθυγράμμιση απόψεων, ευχαρίστως να το εξτάσουμε. Εσείς θα πρέπει να μας υποβάλλετε το αίτημα και θα σας δώσουμε όλο το χρόνο για να μπορέσει να αποφασιστεί από την Επιτροπή. Αυτό είχε συζητηθεί από τους συντονιστές. Θα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν τις κάρτες ψηφοφορίας εάν είναι η ε, σωστή διαδικασία. Συμφωνείτε κύριε Σουάπ και κυρία Γκέπχαρτ να ψηφίσουμε ως χειρός προς το παρόν ή κατευθείαν με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Η ε, πρώτη τροπολογία υπερψηφίσει και ως χειρός και ε, καταπίπτει η τροπολογία 68. Ε, ε, πέρασε και η τροπολογία 16, η τροπολογία 69. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 17 είναι γλωσσικό, δεν θα ψηφιστεί. Τώρα έχουμε την ε, προφορική τροπολογία του κυρίου Κάρας για τους ε, μεμονωμένους τελικούς καταναλωτές υπέρ κατά. Εγκρίνεται. Οπότε οι ράφτες στην Ευρώπη θα ανακουφιστούν. Τροπολογία 18. Είναι επίσης γλωσσολογική 19. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Άρα η 70 καταπίπτει της κυρίας Ρόιτοβα, η 71 επίσης καταπίπτει γιατί καλύπτεται από τη 19, 20 του εισηγητή, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Το άρθρο 4, τροπολογία 72, ε, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 21 καταπίπτει 73 της κυρίας Κόμι Μάντερ Σαλτεμόζερ υπέρ κατά εγκρίνεται άρθρο 5 τροπολογία 22 του εισηγητή Μάντερ υπέρ κατά εγκρίνεται το άρθρο 6 η ε, αίτηση για νέες ίνες Έχουμε μία τροπολογία του κυρίου Μάντες και ε, προφορική τροπολογία που υπάρχει στο κατάλογό σας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 23 καταπίπτει 74 πρόταση σε σχέση με το άρθρο 9 θα ψηφίσουμε ύστερότερα άρθρο 7 τροπολογία 75 αποσύρθηκε τροπολογία 24 μάντες υπέρ κατά εγκρίνεται 25 μάντες υπέρ κατά εγκρίθηκε άρθρο 8 τοπολογία 76 μάντες υπέρ κατά εγκρίθηκε 26 καταπίπτη άρθρο 9 συμβαστική τροπολογία 1 ψηφίζουμε τη συμβιβαστική 1 υπέρ κατά εγκρίθηκε με την έγκριση της συμβιβαστικής τροπολογίας 1 όλες οι άλλες τροπολογίες σε σχέση με αυτό το άρθρο καταπίπτουν και περνάμε τώρα στην τροπολογία 79 Μάντερς υπέρ κατά εγκρίθηκε άρθρο 11 συμβαστική τροπολογία 2 Μάντερς υπέρ κατά εγκρίθηκε. η τροπολογία 29 και 80 καταπίπτουν και περνάμε στη συνέχεια στην τροπολογία 30 μάντες υπέρ. Κατά εγκρίθηκε. Τροπολογία 31 μάντες υπέρ. Κατά εγκρίθηκε. Τώρα περνάμε στη συμβαστική 3. Συμβαστική τροπολογία 3. Υπέρ της συμβαστικής 3. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Τώρα οι τροπολογίες 82 και 81 καταπίπτουν και περνάμε στην τροπολογία 83. Περνάμε στην 83 λοιπόν. Υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 84 υπέρ κατά εγκρίθηκε. Τροπολογία 85 υπέρ κατά εγκρίθηκε αυτή. Η ομάδα της γραμματείας μου μου ανέφερε ενημερωτικά σας το αναφέρω ότι αλλά επειδή αλλάζει η εμβέλεια στην πρόταση θα υπάρξει τεχνική προσαρμογή στο άρθρο 1 της πρότασης που θα γίνει για το τελικό κείμενο όταν επανέλθει. Στο άρθρο 12 η τροπολογία 32 έχει διευθετηθεί, είναι τεχνική, τεχνική προσαρμογή. Περνάμε στην συμβαστική 4 υπέρ κατά εγκρίθηκε. Οι τροπολογίες 33 και 86 καταπίπτουν. Περνάμε στην 34 μάντερς υπέρ κατά. Μπορούμε να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Τροπολογία 34 μάντερς. Άρχεται είπαμε. Άρχεται η ψηφοφορία επί της 34. Τέλος ψηφοφορίας. με μία ψήφο διαφορά καταψηφίστηκε. Αυτό σημαίνει ότι θα περάσουμε στην 87 τώρα τροπολογία. <clears throat> Μακλάκιν. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε την 87 της κυρίας Μακλάκιν. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας καταψηφίστηκε με 5 ψήφους διαφορά, 20 εναντίον, 15 υπέρ. Και περνάμε στην τροπολογία 35, μάντες τώρα. Υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. τροπολογία 88 και 89 καταπίπτουν. Τροπολογία 90, μάντες υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 91 Αρκετά μέλη έχουν προσυπογράψει. Όσοι είναι υπέρ, κατά, καταψηφίστηκε. Τροπολογία 36, Μάντες. Υπέρ, κατά, εγκρίθηκε αυτή. Είμαστε στο κεφάλαιο 3, τίτλο, στον τίτλο. Τροπολογία 37, Μάντες, υπέρ, κατά, εγκρίθηκε. Άρθρο 16, τροπολογία 38, για διαγραφή του κ. Μάντες υπέρ κατά εγκρίθηκε. Άρθρο 17. Εποπτεία αγορά. Τροπολογία 39. Μάντες υπέρ κατά εγκρίθηκε. Τροπολογία 40. Μάντες υπέρ κατά εγκρίθηκε. Τροπολογία 41. 41. Μάντες υπέρ κατά εγκρίθηκε. Τροπολογία 92 του κ. Πουπάκη υπέρ. Ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε. Λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά στην τροπολογία 92. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. 20 υπέρ 17 εναντίον. Εγκρίθηκε. Λοιπόν, η τροπολογία 42 του εισηγητή καταπίπτει. Τροπολογία 43. Μάντερ υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 44. Μάντερ υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. Άρθρο 19 τώρα. Τροπολογία 45. Μάντερ υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 46. Μάντερ υπέρ. Κατά εγκρίθηκε. Τροπολογία 47 όπως έχετε στον πίνακα με την τεχνική μορφή τροπολογία για την πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου υπέρ παρακαλώ κατά εγκρίθηκε η 47 πίτη. 48 του εισηγητή μάντας υπέρ κατά εγκρίθηκε με συγχωρείτε 49 στο άρθρο 20 Μάντερς. υπέρ κατά εγκρίθηκε. Περνάμε στο συμβιβασμό 5, συμβαστική τροπολογία 5, υπέρ του συμβιβασμού 5, κατά εγκρίθηκε. Τώρα λοιπόν έτσι θα περάσουμε οι 50 και οι 93 καταπίπτουν. Περνάμε στην 51 μάντερς υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Η τροπολογία 95 λοιπόν καταπίπτει σαν συνέπεια τούτου άρθρο 21α νέο προσωρινά μέτρα. Συμβαστική τροπολογία 6 υπέρ κατά εγκρίθηκε έτσι 52 και 96 καταπίπτουν περνάμε στην τροπολογία 53 μάντερς υπέρ κατά εγκρίθηκε τροπολογία 54 μάντερς υπέρ κατά και αυτή εγκρίθηκε. Παράρτημα 5. Τροπολογία 97. Στην 97 ηλεκτρονική ψηφοφορία άρχεται η ψηφοφορία από τις 97. Πέρας ψηφοφορίας καταψηφίστηκε 18 εναντίον 17 υπέρ. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 98. 98. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά επί της 98. Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα καταψηφίστηκε και αυτή. 15 υπέρ 17 εναντίον. Περνάμε στην τροπολογία 55. Μάντες. Υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 99 υπέρ κατά απορρίφθηκε τώρα η τροπολογία 100 κ. Καράς καταπίπτει και αυτή περνάμε τώρα στις αιτιολογικές σκέψεις τροπολογία 1 Μάντερσε υπέρ κατά εγκρίθηκε τροπολογία 2 του εισηγητή υπέρ κατά εγκρίθηκε τροπολογία 3 υπέρ κατά εγκρίθηκε τροπολογία 4 υπέρ κατά εγκρίθηκε τροπολογία 5 υπέρ κατά εγκρίθηκε τροπολογία 6 υπέρ κατά εγκρίθηκε τροπολογία 57 υπέρ κατά εγκρίθηκε η τροπολογία 7 και η 58 καταπίπτουν τροπολογία 8 μάντερς υπέρ κατά εγκρίνεται Τοπολογία 59, Ρόιτοβα, υπέρ. Κατά, εγκρίθηκε. Η 9 αποσύρθηκε. Τροπολογία 10, Μάντες, υπέρ. Κατά, εγκρίθηκε. Τροπολογία 11, Μάντες, υπέρ. Κατά, εγκρίθηκε. Η τροπολογία 60 καταπίπτει. Περνάμε στη συμβαστική τροπολογία 7 για την αιτιολογική σκέψη υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Οι 61, 62 και 67 καταπίπτουν όλες. Περνάμε στην 63 τροπολογία. υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. Οι 12 καταπίπτει λοιπόν. Περνάμε στο συμβιβασμό 8. Υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. Και έτσι οι 13, 64, 65, 66 καταπίπτουν όλες. Περνάμε στην αιτιολογική σκέψη για την 20 τώρα. Υπέρ. Κατά εγκρίθηκε. Και τώρα πάμε και ψηφίζουμε το σχέδιο έκθεσης με ηλεκτρονική ψηφοφορία όμως. Άρχεται η ψηφοφορία επί του σχεδίου έκθεσης παρακαλώ. Ψηφοφορία ηλεκτρονική επί του σχεδίου έκθεσης. Άρχεται. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε λοιπόν. 37 συμμετείχαν, 30 υπέρ, ένας εναντίον, 6 αποχές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ Σιγητά. Έχετε κάποιες τελικές παρατηρήσεις. Πολύ καλά. Για το Συμβούλιο και την Επιτροπή κάποια σχόλια, όχι σε αυτή τη φάση. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας. Περνάμε λοιπόν τώρα στην ψήφιση της έκθεσης Στάιλερ. Πού είναι η κυρία Στάιλερ, εδώ είναι. Α, έχετε καθίσει σε άλλη θέση. Ωραία. Θα θέλατε ίσως να κάνετε εισαγωγικά κάποιες παρατηρήσεις για την έκθεσή σας πριν ψηφίσουμε για την γνωμοδότηση. Uh, uh, Ευχαριστώ. Δεν έχω κάτι να προσθέσω. Μπορούμε να περάσουμε απευθείας στις ψηφοφορίες, αλλά θα ήθελα να ευχαριστήσω τους σκιώδεις συζητητέ και όσους ε, κατέθεσαν τροπολογίες νομίζω ότι βοήθησαν την έκθεση. Περιμένω με ανυπομονησία την ψηφοφορία. Πολύ ωραία. Ας περάσουμε στην ψηφοφορία για την έκθεση Στάιλερ. Παραγραφός 1. Τροπολογία 2. Στάιλερ Λεγκρίπ. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία Σφένσον. Προσθήκη. Υπέρ. Ακαλύτερα να το κάνουμε ηλεκτρονικά. έναρξη ψηφοφορία για την τροπολογία Σφένσον. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 20 υπέρ 15 κατά. Μετά τροπολογία 3 Νικουλέσκου. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 4 Σβένσον. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 5. Λεγκρίπ. Έναρξη ψηφοφορίας ηλεκτρονικά. Τροπολογία 5 Λεγκρίπ. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 21 ψηφί υπέρ, 15 κατά. Τροπολογία 6, Νικουλέσκου, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Μετά, η κυρία Γκρίπ προτείνει προφορική τροπολογία που βλέπετε στον κατάλογο. Συμφωνείτε κυρία Στάιλερ. Υπέρ της προφορικής τροπολογίας. Κατά εγκρίνεται. Άρα καταπίπτει η αρχική τροπολογία Λεγκρίπ, τροπολογία 7 Νικουλέσκου υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Σφένσον 9 υπέρ. Κατά. Να το εξετάσουμε. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Έναρξη ψηφοφορίας. Τροπολογία 9 Σφένσον. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 23 ψήφοι υπέρ, 14 κατά. Περνάμε στην τροπολογία 10. Λεγκρίπ. Ηλεκτρονικά. Ψηφοφορία για την τροπολογία 10. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 22 υπέρ, 13 κατά, 2 αποχές. Τροπολογία 11 υπέρ. Και εδώ ηλεκτρονικά. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας ψηφοφορίας. 18 υπέρ 18 κατά, κατά απορρίπτεται, με συγχωρείτε. Τροπολογία 12 Νικουλέσκου. Υπέρ κατά εγκρίνεται 13 Στάιλερ υπέρ κατά εγκρίνεται 14 Νικουλέσκου υπέρ κατά εγκρίνεται 15 Λεγκρίπ υπέρ κατά εγκρίνεται 16 Λεγκρίπ Σουβάν υπέρ κατά εγκρίνεται 17 υπέρ κατά εγκρίνεται. Έναρξη ψηφοφορίας για το σχέδιο γνωμοδότησης στο σύνολό της. Έναρξη ψηφοφορίας παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 30 ψήφοι υπέρ και 6 αποχές. Σας ευχαριστούμε κυρία Στάιλερ και πιστεύω ότι θα συνεργαστείτε και θα εργαστείτε σκληρά για να συμπεριληφθούν οι τροπολογίες μας στην ψηφοφορία της Επιτροπής Βιομηχανίας. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας και αυτό που προτείνω να κάνουμε τώρα είναι να συνεχίσουμε τη συζήτηση για την έκθεση Γκρέχη. Ζητήσαμε από τον κύριο Μόντι να επανέλθει στις 11 για την ομιλία του. Οπότε κάποιοι ίσως θα έρθουν εκείνη την ώρα. Για να δούμε λοιπόν ποιοι είναι οι ομιλητές που παραβρέσκονται ήδη εδώ. Αν και βεβαίως κάποιοι μπορεί να θέλουν να επανέλθουν μετά τον κύριο Μόντι. Αν κάποιος άλλος θέλει να συμπεριληφθεί, ενδεχομένως και άλλοι εργαζόμενοι εισηγητές σε θέματα εσωτερικής αγοράς, παρακαλώ μπορούμε να σας συμπεριλάβουμε στον κατάλογο μιλητών. Έχουμε αρκετό χρόνο για συζήτηση. Ο κύριος Τριανταφυλλίδης ήδη ενδιαφέρθηκε. Ελπίζω και κάποιοι άλλοι από εσάς να συμμετέχουν στη συζήτηση. Το λόγο έχει η κυρία Γκέπχαρτ. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ επίσης τον Λουί Γκρέκ για την πραγματικά πολύ καλή δουλειά που έκανε. Είναι μια πάρα πολύ καλή έκθεση αυτή που και πάρα πολλά σημαντικά σημεία συμπεριλαμβάνει που νομίζω για τους πολίτες γυναίκες και άντρες της Ένωσης και για τους καταναλωτές έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Λοιπόν, θα ήθελα σε ένα σημείο να αναφερθώ που νομίζω ότι και από διαφόρους προαναφέρθηκε, αλλά είναι σημαντικό και αυτό το σημείο. Δηλαδή να δώσουμε μια απάντηση. Πώς μπορούμε τους πολίτες μας να τους ξανακερδίσουμε πάλι για την Ευρώπη, υπέρ της Ευρώπης, υπέρ της σκέψης για την ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την απογοήτευσή τους, να ξεπεράσουμε τη δυσφορία τους. Είναι νομίζω ένα από τα μεγάλα ε, έργα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και νομίζω ότι η σωστή αντιμετώπιση εξευρίσκεται. Για εκείνου που ανέφεραν ότι πολλά σημεία βρίσκουν ότι λείπουν σε αυτή την έκθεση θα ήθελα να του πω ότι αφενό. Ο κύριος Γκρέκ δεν είχε περισσότερο χώρο για να συντάξει ευρύτερο, σε ευρύτερο πλαίσιο αυτή την έκθεση και πολλές προτάσεις που προαναφέρθηκαν δεν εμπίπτουν υποχρεωτικά μέσα σε αυτό το πεδίο στο οποίο αναφέρεται η έκθεση Γκρέκ. Να αναφέρω για άλλη μια φορά την έκθεση δημιουργία μιας εσωτερικής αγοράς για τους ε, καταναλωτές και τα δικαιώματα των καταναλωτών και των πολιτών. Είναι σημαντικό τέτοιου είδους θέματα όπως πνευματική ιδιοκτησία, intellectual property είναι σημαντικά, αλλά δεν είναι αυτά τα οποία είναι για τους καταναλωτές τα πιο σημαντικά. Έτσι. Είναι κάπως περισσότερο αυτά για την Ευρώπη των ε, επιχειρηματιών και της εσωτερικής αγοράς. Πρέπει να κάνουμε μια σωστή επιλογή πιστεύω όταν έχουμε έναν αντίστοιχο τίτλο. Τι θέλουμε να εντάξουμε σε αυτό τον τίτλο, σε αυτό το πλαίσιο. Πώς θα θέσουμε τις προτεραιότητες. Ή και ίσως κάποιοι επιθυμούν να έχουμε μια ευρύτατη συζήτηση όλα επί, του επιστητού, επί παντός του επιστητού να ενταχθούν όμως το πολιτικό μήνυμα τι θα γίνει έτσι υπονομεύεται, δεν μπορεί να περάσει. Είναι το θέμα το οποίο μέσα σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να δούμε και να θέσουμε αυτό το ερώτημα στους εαυτούς μας και να συζητήσουμε για αυτά τα πράγματα. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι αυτά τα θέματα δεν είναι σημαντικά. Όχι, δεν θέλω να πω ότι δεν είναι σημαντικά. Είναι όμως τίθεται το θέμα πώς θα θέσουμε κέντρα βάρους και προτεραιότητες σε αυτή την έκθεση. Και γι' αυτό πιστεύω ότι ο κύριος Γκρέκ, ο Λουί Γκρέκ, πολύ σωστά έκανε τις σωστές επιλογές επιλέγοντας αυτά τα στοιχεία ως προτεραιότητες. Αυτό ανταποκρίνεται και στην εντολή που εμείς ως συντονιστές, ως Επιτροπή δώσαμε στο Λουί Γκρέκ τη δημιουργία <clears throat> μιας εσωτερική αγοράς για τους καταναλωτές και τους πολίτες. Αυτό είναι το πρώτο που θέμα αρχή θα ήθελα να θέσω και να αποσαφηνίσω. Το δεύτερο στη συνέχεια. Και νομίζω και αυτό είναι πολύ σημαντικό και σωστά πρέπει να μπορεί να περάσει από την πρόταση του Λουίς και σωστά περνάει. Είναι αυτό λοιπόν το ότι εμείς πρέπει να προσδιορίσουμε εκ νέου πώς θα αντιμετωπίσουμε στη συνέχεια την εσωτερική αγορά. Τι ανήκει σε αυτή την εσωτερική αγορά από την ιστορική εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απορρέει και είναι σημαντικό ότι η επιχειρηματική πολιτική, η χρηματοοικονομική πολιτική ήταν πάντα στο προσκήνιο περισσότερο. Και πολλοί πολίτε διαρωτώνται πού βρισκόμαστε εμεί ω πολίτε, πού βρισκόμαστε εμεί ω καταναλωτέ, οι εργαζόμενοι, οι πολίτε, πού βρίσκονται, πού βρισκόμαστε, ποια αξία και ε, σημασία έχουμε. Και με τι συνθήκε τη Αβώνα έχουμε τώρα πια μια νέα δυνατότητα να δράσουμε ω θέμα αρχή πλέον. Και από αυτού ο Λουί Γκρέκα σωστά αντιμετωπίζει τα θέματα στην έκθεσή του. Έτσι στο άρθρο 3 και στο άρθρο 4, στο 7, στο 9, 14 <clears throat> της συνθήκης αυτά που συμπεριλαμβάνονται αφενός όσον αφορά την οικονομία, κοινωνική οικονομία της αγοράς και τα κοινωνικά θέματα αφενός, αφετέρου αυτά τα οποία συνδέονται με αυτή την πτυχή. Δηλαδή ότι τα δικαιώματα των καταναλωτών γυναικών και ανδρών έχουν μια οριζόντια πλέον εγκάρσια διάσταση και προοπτική. <clears throat> η προστασία των καταναλωτών προωθείται μέσω της συνθήκης Λισαβόνας έτσι. Και έτσι πρέπει να ε, βρεθούμε στο ύψος των περιστάσεων να ανταποκριθούμε σε αυτή την πραγματικότητα. Και πολύ καλά νομίζω το εκπονεί ο Λουί Γκρέκ στην έκθεση που έχουμε μπροστά μας. Το τρίτο σημείο, όπου και σε αυτό πάλι πρέπει, μπορούμε να εγγράψουμε στα λάβαρά μας στις σημαίες μας ε, ως κοινοβούλιο και αυτό το οποίο έχει συντάξει εδώ Λουί τι είναι. Είναι το ότι η ενιαία εσωτερική αγορά δεν είναι αυτός σκοπός. Δεν είναι ομφαλοσκόπηση, είναι σημαντικό και αυτό να το διαπιστώσουμε. Δεν είναι αυτό σκοπός λοιπόν. Είναι ένα μέσο για την επίτευξη ενός στόχου. Είναι ένα εργαλείο και έτσι εμείς πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, να δραχθούμε τις ευκαιρίες χρησιμοποιώντας αυτό το μέσο, αυτό το εργαλείο για να πετύχουμε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη από πλευράς των πολιτών στην Ένωση, σε αυτά που κάνουμε. Αυτή είναι μια έννοια που θα ήθελα ευχαρίστως να προτείνω στον ε, Λουί. Ε, στο Λουί Γκρέκ. Δηλαδή η εμπιστοσύνη των πολιτών πιο έντονα, πιο ενισχυμένα να μπορέσει να ενταχθεί σε αυτήν την έκθεση. Ότι πρέπει να μεριμνήσουμε η εμπιστοσύνη των πολιτών στην εσωτερική αγορά να ενδυναμωθεί, να ενισχυθεί. Και γι' αυτόν τον λόγο εμεί πρέπει πιο ενισχυμένα να τονίσουμε εμεί εδώ ότι η εσωτερική αγορά είναι κάτι παραπάνω από την οικονομία, κάτι παραπάνω από τα χρηματοοικονομικά θέματα. Είναι προστασία καταναλωτών, είναι κοινωνικά δικαιώματα και οικολογικά δικαιώματα. Έχει απόλυτο δίκιο γι' αυτό η κυρία Ρούιλε αλλά και αυτό αναφέρεται και στην έκθεση του Λουί. Αλλά θα θέλαμε να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο αν γίνεται, παρακαλώ. Και μετά για τα θέματα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Και αυτά εντάσσονται στην έκθεση του Λουί Γκρέκ. Το χαιρετίζω όμως ότι δεν έχουν την ανώτατη ε, έσχατη προτεραιότητα, διότι είναι ένα θέμα το οποίο βρίσκεται πολύ έντονα συζήτηση αυτή τη στιγμή. Και είναι σωστό να ε, συζητείται έντονα σε αυτή τη συγκυρία. Τα δικαιώματα των καταναλωτών σε αυτό τον τομέα πρέπει να ενισχυθούν και σημαντικά κιόλα. Όμω ο φόβο τη ομάδα μα ως σοσιαλιστών είναι αν αυτά τεθούν στο προσκήνιο, όλοι οι άλλοι τομεί θα απομονωθούν, θα ε, ξεχωριστούν και θα ξεχαστούν, θα αμεληθούν. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι πολύ ευρύτερο όμω από την άλλη πλευρά από το να συζητάμε μόνο για τι χρηματικέ υπηρεσίε που είναι μεν πάρα πολύ σημαντικές <clears throat> γιατί πρέπει να υπάρξει η εμπιστοσύνη των πολιτών με σαφείς κανόνες που θα δημιουργήσουμε για τα χρηματικά τα οικονομικά θέματα. Όμω, ο άλλο τομέα για την αποκατάσταση τη εμπιστοσύνη των πολιτών, οι ευρύτερε άλλε πτυχέ είναι και αυτέ εξίσου σημαντικέ. Ένα άλλο τελευταίο στοιχείο που θα ήθελα να αναφέρω, παρότι υπάρχουν πάρα πολλά περισσότερα ακόμα, είναι ο τομέα που επιμέρου αναφέρθηκε από κάποιου συναδέλφου, Δηλαδή το θέμα της δημιουργίας ενός νομικού πλαισίου για την παροχή υπηρεσιών στη γενικού οικονομικού συμφέροντος κοινού ωφέλους. Και νομίζω ότι ένα από τα συμπεράσματα ακριβώς που και εγώ για την ομάδα μου θέλω να ξανατονίσω για άλλη μια φορά από αυτή τη συζήτηση για, για την ε, οδηγία περί παροχής υπηρεσιών, ένα σημαντικό συμπέρασμα. Είχαμε μια έντονη συζήτηση στην οδηγία περί υπηρεσιών και εδώ στην Ευρωβουλή και στο Συμβούλιο. Αν αυτές οι υπηρεσίες ανήκουν στην οδηγία περί παροχής υπηρεσιών ή όχι οι υπηρεσίες ολικού συμφέροντος. Είναι εμπορικής μορφής ε, υπηρεσία ή όχι ή μήπως δεν είναι εμπορικές, εμπορικού χαρακτήρα υπηρεσίας. Και είπαν και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεν είναι κανονικές ε, ε, υπηρεσίε που εντάσσονται ή που μπορούν να ενταχθούν στην οδηγία περί υπηρεσιών. Ξεχωριστά πρέπει να αντιμετωπιστούν αυτέ. Και αυτό γιατί. Διότι οι συνθήκε πλαίσιο που διαμορφώνουν αυτέ είναι πολύ διαφορετικέ. Δεν πρόκειται μόνο για δικαίωμα καταναλωτών αλλά και δικαιώματα ασθενών για παράδειγμα και για τι κοινωνικέ υπηρεσίε και για τα δικαιώματα εδώ επιπλέον των πολιτών εκείνων που βρίσκονται σε ιδιαίτερη ανάγκη και έχουν ιδιαίτερες ανάγκες. Πρέπει οι ειδικές αυτές ανάγκες να ληφθούν υπόψη. Πρόκειται για καθολικές, καθολικούς συμφέροντος υπηρεσίες που έχουν ιδιαίτερη σημασία και είναι ξεχωριστές. Αυτό είναι εκείνο το οποίο <clears throat> αποφασίσαμε να γίνει. Και γι' αυτό το συμπέρασμα ακριβώς είναι το σωστό συμπέρασμα. Να πει δηλαδή κανείς ότι δεν μπορούμε να αγνοήσουμε αυτά τα θέματα και να μην δώσουμε συνέχεια, διότι η συνθήκη της Λισαβόνας με το άρθρο 14 και το πρωτόκολλο για αυτό το θέμα δίνει εντολή σε μας να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα στη συνέχεια και να δώσουμε συνέχεια και να μην το αφήσουμε <clears throat> στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, στο 10 Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή και σε άλλους που αναπερίπτωση θα λένε τι πρέπει να γίνει επιμέρους. Εμείς πρέπει να εξετάσουμε και να δούμε ποια συνέχεια θα δώσουμε σε αυτά τα θέματα. Και όταν λέει ο Λουί Γκρέκ ότι χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο για αυτόν τον τομέα και ίσως σε διαπραγματεύσεις με τους συναδέλφους που είπαν ότι έχουν κάποιους φόβους ότι θα υπάρξει γραφειοκρατική επιβάρυνση και ότι ουσιαστικά ίσως ανήκει στην, ε, σε σχέση με τις παρεμβάσεις για την επικουρικότητα πρέπει να αποσαφηνίσουμε ότι εδώ αυτό περί το πρόκειται είναι η προστασία αυτών των υπηρεσιών που πρέπει να διασφαλιστεί ώστε να παραμείνουν στα κράτη-μέλη ως υπηρεσίες σύμφωνα με τις ανάγκες των πολιτών επιτόπου στις, στα κράτη-μέλη και να διαμορφώνονται ανάλογα με τις ανάγκες των πολιτών χωρίς να υπάρχουν φόβοι όσον αφορά κυβερνήσεις ή αρχές το τι θα πρέπει να γίνει επειδή δεν θα υπάρχει κάποιο δεδομένο νομικό πλαίσιο για αυτόν τον τομέα. Γι' αυτό πρέπει πολύ εξειδικευμένα να συζητήσουμε χειροπιαστά για αυτό το θέμα. Να μην το αμελήσουμε ή το αναβάλουμε. Να δούμε πώ μπορεί να δημιουργηθεί ένα τέτοιο πλαίσιο ώστε οι φόβοι που εκφράστηκαν σε σχέση με αυτά πιο πριν να μπορούν να ληφθούν υπόψη και να αντιμετωπιστούν, να ξεπεραστούν. Ακριβώ ε, όσα είπε η κυρία Ρούιλε και ο κύριο Σβάμπ για αυτό το θέμα. Για να μπορέσουμε να τα κανονίσουμε σωστά τα πράγματα. Δεν πρόκειται για εμπορικές υπηρεσίες ή για αντικείμενα προς εμπορική εκμετάλλευση, αλλά το αντίθετο για την προστασία τους. Να διαμορφώσουμε πλαίσια προστασία ε, προστασίας αυτών των υπηρεσιών. Αυτό κατανόησα και αυτά ήθελα να πω μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Και μακρηγόρησα ίσως κάπως, διότι <clears throat> είπε ο πρόεδρος στην αρχή της συζήτησης ότι σήμερα έχουμε παρκή χρόνο λέει, πολύ χρόνο και έτσι πήρα, α το πω έτσι, το δικαίωμα, αυθερέτησα, ώστε να μακρηγορήσω λίγο περισσότερο γι' αυτό. Ευχαριστώ. Ναι, αλλά ήταν πολύ καλή η παρέμβασή σας και όπως είπα για αυτή την πολύ σημαντική έκθεση έχουμε φροντίσει να έχουμε πολύ χρόνο για τη συζήτηση. Θα περιμένουμε μέχρι τις 11 για την ομιλία του κυρίου Μόντι γιατί έχουμε και web streaming και δεν ξέρω μπορεί να περιμένουν πολλά μέσα ενημέρωσης για να τον ακούσουν χωρίς να θέλω και να αυξήσω ιδιαίτερα τις ελπίδες σας. Ίσως όμως να με παρακολουθεί ο συνάδελφος για να καταλάβει πώς ακριβώς λειτουργούμε στην εσωτερική αγορά. Να πω σε όλους τους συναδέλφους που είναι γραμμένοι στον κατάλογο ότι όλοι θα έχουν χρόνο να μιλήσουν και να σχολιάσουν και τα όσα θα πει ο κύριος Μόντι. Και με συγχωρείτε που δεν το είπα προηγουμένως, αλλά έχουμε μία νέα συνάδελφο, Γαλίδα, την κυρία Σουλή και το λόγο έχει η κυρία Στάιλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομη καθώς πολλά θέματα έχουν ήδη αναφερθεί. Σκεφτόμουν ότι όταν μιλάμε για την εσωτερική αγορά και έχουμε και την επιτροπή μας που είναι Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς μπορεί να προκύψουν συγχύσεις. Ίσως θα έπρεπε να το σκεφτούμε λίγο γιατί μερικές φορές Μιλάμε για εσωτερική αγορά και αυτό ακούγεται ως ε, προστατευτισμός σε αντίθεση με την ενιαία αγορά. Ίσως θα έπρεπε να το σκεφτούμε και για το όνομα της Επιτροπής μας. Θα ήθελα να πω ότι για το 8, όσον αφορά δηλαδή τους 20 ε, μεγαλύτερους λόγους απογοητεύσης από την ε, εσωτερική αγορά καλός, αλλά ίσως θα έπρεπε να ασχοληθούμε με τα τρία βασικότερα ή τα πέντε βασικότερα, να είμαστε δηλαδή πιο συγκεκριμένοι και πιο επιθετικοί για τα συγκεκριμένα αυτά θέματα. Επίσης, χαιρόμαι που αναφέρεστε στο Solvit, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Το ανέφερα και ο Πρόεδρος και άλλοι, όμως είναι σημαντικό να έχουν έναν τρόπο οι πολίτες να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Το συζητήσαμε και στην ομάδα εργασίας. Πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν τι ακριβώς είναι η εσωτερική αγορά και τι ωφέλη περιέχει για αυτούς. Γι' αυτό χαίρομαι που βρίσκεται και σήμερα μαζί μας ο κύριος Μόντι, γιατί φαίνεται πόσο σημαντικό είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε, αλλά και πόσο ενδιαφερόμαστε για αυτό που κάνετε εσείς. Αναμένουμε λοιπόν με ανυπομονησία την έκθεσή σας. Όσον αφορά τώρα τον χάρτη των πολιτών, είναι ενδιαφέρον όμως, αν πρόκειται να κάνουμε κάτι τέτοιο, πρέπει να παραμείνει πολύ απλό και να ενημερώνει τους πολίτες για τα δικαιώματά τους. Με βάση την συζήτηση που είχαμε και χτες αλλά και σήμερα φαίνεται ότι όντως πρέπει να κάνουμε κάτι γι' αυτό γιατί η ενιαία αγορά είναι ίσως το σημαντικότερο κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν δεν λειτουργεί σωστά τότε αυτό πλήττει όλους μας. Σας ευχαριστώ για τη συζήτηση και αναμένω τις 11 η ώρα όπου θα ξεκινήσει να μιλάει ο κύριος Μόντι. Ευχαριστώ. Κυρία Τούρμ. Thank you. Um, this, this is uh, really... Ευχαριστώ. Είναι συζήτηση βάσης αυτή και είναι ενδιαφέρον που έχουμε τέτοιου είδου συζήτηση στην Επιτροπή μας που ορισμένες φορές ασχολείται με πολύ τεχνικά και συγκεκριμένα θέματα. Χαίρομαι λοιπόν που έχουμε μια συζήτηση για την κατεύθυνση της εσωτερικής αγοράς συμφωνώ με την κυρία Κέιπχαρτ ότι η εσωτερική αγορά δεν πρέπει να είναι αυτός σκοπός. Είναι εργαλείο για να έχουμε ισχυρότερες οικονομίες και για να χρηματοδοτήσουμε πολύ φιλόδοξες κοινωνικές αγορές και περιβαλλοντικές αλλαγές. Πρέπει λοιπόν να το θυμόμαστε. Είναι εργαλείο προκειμένου να αποκτήσουμε μία βιώσιμη αηφόρο κοινωνία. Είναι μεν η εσωτερική αγορά αυτή τη στιγμή ατμομηχανή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, αλλά δεν έχουμε καταφέρει να έχουμε μια ολιστική προσέγγιση που θα συμπεριλαμβάνει και άλλες διαστάσεις όπως η περιβαλλοντική. Γι' αυτό χαίρομαι που βλέπω την έκθεση να τονίζει τα προβλήματα που υπάρχουν. Γιατί τα προβλήματα δεν είναι μόνο η εφαρμογή και η γραφειοκρατία, αλλά και το κοινωνικό ντάμπιν, ο αθέμητος ανταγωνισμός, οι συνθήκες εργασίας, η φοροδιαφυγή κτλ. Γιατί αν δεν τα αντιμετωπίσουμε αυτά, τότε ποτέ δεν θα καταφέρουμε τους ανθρώπους να ερωτευθούν την Ευρώπη. Χρειαζόμαστε λοιπόν περισσότερη ολοκλήρωση, ολοκλήρωση της αγοράς. Αλλά για να γίνει αυτό θα χρειαστούν κάποιες σημαντικές προϋποθέσεις. Καταρχάς, αποτελέσματα για τους καταναλωτές. Αυτό το καλύπτει πολύ καλά η έκθεση. Επίσης, διαφάνεια, σαφή και υψηλά δικαιώματα. Επίσης, Καλό είναι που έχουμε μία λίστα με τα προβλήματα που μας απογοητεύουν, αλλά ίσως θα χρειαζόμασταν και ένα κατάλογο με τα καλά, με αυτά που είναι σωστά και θετικά στην εσωτερική αγορά. Επίσης, κάποιες προϋποθέσεις για τη μείωση του αθέμητου ανταγωνισμού, που θα χρειαζόταν πολύ ευρέα μέτρα. Πρέπει να δούμε θέματα όπως η φορολόγηση επιχειρήσεων, συνθήκες εργασίας και οι προϋποθέσεις που ισχύουν όσον αφορά το κλίμα. και νομίζω ότι στις ε, παραγράφους 26, 50 και 52 αναφέρονται αυτά τα θέματα αλλά καλό θα ήταν να τα τονίσουμε ακόμη περισσότερο. Τέλος, να πω ότι αυτή η συζήτηση μας δείχνει το δρόμο και προς μία ακόμη πιο ευρεία συζήτηση όσον αφορά το πρόβλημα με τη σύγχυση στις αρμοδιότητες. Έχουμε πολλές αρμοδιότητες, αλλά συχνά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι σε θέματα κοινωνικά ή περιβαλλοντικά και δυστυχώς αυτό το πρόβλημα της σύγχυσης δεν έχει επιληθεί ακόμη. Έχουμε τη νέα συνθήκη βεβαίως και πρέπει να ακολουθούμε τις γραμμές της συνθήκες, αλλά ίσως θα έπρεπε για την επόμενη... Δεν τολμώ καν να το πω, αλλά εν πάση περιπτώσει για την επόμενη συνθήκη ίσως θα έπρεπε να επαναξετάσουμε το όλο θέμα των αρμοδιοτήτων. Ευχαριστούμε. Η κυρία Ράπτη τώρα και μετά ο κύριος Μόντι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα μιλήσω για αυτή την έκθεση με τα λόγια που μου μιλούν οι ψηφοφόροι μου στην Ελλάδα. καταρχήν είναι ένα, μια, πραγματικά ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και για το παρόν και για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η έκθεση του Λούι το χειρίστηκε εξαιρετικά. Θέλω να τον ευχαριστήσω γι' αυτό ε, ξέρετε η εσωτερική αγορά στα μάτια των ε, ελλήνων πολιτών είναι σαν μια κυρία πάρα πολύ δύσκολη να την καταλάβεις σαν μια κυρία με άσχημο πρόσωπο με πολύ σκληρή καρδιά και πολύ μακριά από τις ανάγκες και την καθημερινότητά τους. νομίζω ότι η εσωτερική αγορά θα πρέπει να αλλάξει πρόσωπο. Ε, είναι χαρακτηριστικό ότι όταν με ρωτούν σε ποια επιτροπή συμμετέχω και απαντώ ότι συμμετέχω στην επιτροπή εσωτερικής αγοράς η απάντηση ε, τις, περισσότερες φορές είναι ένα μ και ένα κούνημα του κεφαλιού τι μας λες τώρα. αυτό νομίζω ότι δεν θέλω να το ξανακούσω και αυτή η έκθεση την οποία χειριζόμαστε τώρα μας δίνει μια πολύ καλή ευκαιρία ε, θέλω η εσωτερική αγορά να γίνει μια κυρία όμορφη με πολύ καλό δυνατό μυαλό αλλά και με μια πολύ δυνατή ψυχή. Όταν μιλάω για μυαλό και για ψυχή καταλαβαίνετε όλοι σας ότι μιλάω για την οικονομική ματιά και για την κοινωνική ματιά που πρέπει να έχει η εσωτερική αγορά θεωρώ ότι η εσωτερική αγορά όπως πολύ καλά είπε και με κάλυψε απολύτως η εύελιν και η συνάδελφος η έμιλι τουρούνεν δεν υπάρχει μόνο και μόνο για τα χαρτιά. η εσωτερική αγορά θεωρώ ότι υπάρχει για τους πολλούς και ευάλωτους πολίτες και όχι για τους λίγους και ισχυρούς. έτσι λοιπόν εστιάζω σε ένα σημείο από τα πολλά τα οποία χειρίζεται ο Λούις στην έκθεσή του στο θέμα των καταναλωτών και των πολιτών. νομίζω ότι για να προοδεύσει και να αναπτυχθεί η εσωτερική αγορά χρειάζεται την υποστήριξη των πολιτών άρα θα πρέπει να φροντίσει για αυτούς θα πρέπει να φροντίσει για τα δικαιώματά τους ώστε και αυτοί με τη σειρά τους να αγκαλιάσουν την εσωτερική αγορά και να της δώσουν τη θέση που πρέπει και μέσα σε κάθε κράτος μέλος αλλά και μέσα στην καρδιά τους το τελευταίο μπορεί να ακούγεται ρομαντικό αλλά επιμένω ότι δεν είναι γιατί τους πολίτες τους χρειαζόμαστε στην ευρώπη να δουλεύουν για την ευρώπη να στηρίζουν την εσωτερική αγορά. ο ενημερωμένος καταναλωτής θα μπορέσει να διεκδικήσει τα δικαιώματά του να κάνει χρήση της εσωτερικής αγοράς και άρα να βοηθήσει στο να καταπολεμηθούν κακές πρακτικές. είναι ε, από τη μια μεριά δυσνόητα, από την άλλη μεριά όμως και πάρα πολύ εύκολα και απλά τα πράγματα. Ε, καταλήγοντας, νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία η εσωτερική αγορά να γίνει κατανοητή από τους πολίτες. Και επειδή είναι ένας πολύ μεγάλος τομέας που είναι δύσκολο να αισθανθεί κάποιος ότι τον πιάνει αυτό το τομέα στα χέρια του, νομίζω ότι θα πρέπει ε, μια ιδέα, λέω, να επιλεγούν ένα ή δύο θέματα εύκολα σχετικά να τα αντιληφθεί ο καταναλωτής ώστε πραγματικά να δοθούν παραδείγματα στην πράξη. Άκουσα για παράδειγμα από έναν προηγούμενο συνάδελφο, από τον Κούε, αν δεν κάνω λάθος, την ε, υπόθεση των 5 ε, ευρώ που πληρώνουμε περισσότερο ε, στις διατραπεζικές μας συναλλαγές. Ένα παράδειγμα λέω τυχαίο. Θα μπορούσαμε με αυτό να κάνουμε μια καμπάνια ή επιλέγοντας ένα άλλο παράδειγμα να κάνουμε μια καμπάνια και να καταλάβει ο κάθε πολίτης, ο απλός πολίτης ότι η εσωτερική αγορά είναι για το συμφέρον του τον εξυπηρετεί και γι' αυτό θα πρέπει να την υπηρετεί και αυτός. Ε, κλείνω εδώ και πραγματικά εκφράζω την αισιοδοξία μου ε, για την πορεία αυτής της έκθεσης και ευχαριστώ και πάλι τον Λουί. Αλλά πριν κλείσω και ε, για να μην ξαναπάρω το λόγο μετά θα ήθελα να ρωτήσω τον καθηγητή Μόντι τον οποίο ευχαριστώ που είναι εδώ όπως τον ευχαριστώ και για την εισήγηση που είχε κάνει στις 14 Δεκεμβρίου στο Στρασβούργο θα ήθελα να τον ρωτήσω πραγματικά τι θα κάνει για να κάνει την εσωτερική αγορά, τι θα εισηγηθεί για να κάνει την εσωτερική αγορά περισσότερο ελκτική για τους πολίτες και πώς θα μπορέσει να πείσει τους πολίτες ότι το οικονομικό ή κοινωνικό πρόσωπο της Ευρώπης δεν είναι δίλημα, είναι ψεύτο δίλημα. Πώς θα βρούμε δηλαδή μια ισορροπία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Ράπτη. Με εντυπωσίασε η τώρα μάσας της ενιαίας αγοράς και πολύ μου άλλασε η κομψή κυρία με ισχυρό πνεύμα και δυνατή καρδιά. Νομίζω ότι όλες οι κυρίες αυτής της Επιτροπής νομίζω ότι μπορούν να περιγραφούν με τον ίδιο τρόπο. Είναι μια λοιπόν ενδιαφέρουσα εισαγωγή για τον ειδικό προσκαλεσμένος μας τον κύριο Μόντι σήμερα το πρωί που θα μας μιλήσει για την ενιαία αγορά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που με καλέσατε και που μου δώσατε ε, το, το καλύτερο χρόνο από πλευράς της αναμετάδοσης ε, στο διαδίκτυο ε, κατά τρόπον ώστε να κάνω τα σχόλιά μου αν και υποθέτω ότι και εσείς θα κάνατε σχόλια εφόσον η κυρία Ράπτη τόσο ωραία περιέγραψε την ενιαία σαν μία ισχυρή, κομψή και δυναμική παρουσία και εκπροσώπηση σε αυτήν την Επιτροπή. Θα ήθελα να εκφράσω την ε, ε, ε, εκτίμησή μου και το θαυμασμό μου για την έκθεση ε, Γκρέκ και ε, για ε, τον πρόεδρο που αποφάσισε να συνταχθεί μία έκθεση για την ενιαία αγορά στην Επιτροπή σας ένα θέμα το οποίο έχει πολύ σημαντική σημασία πολιτική και γενική και την ποιότητα της εκθέσεως του Λουί που ε, έχει τύχει των επένων όλων ε, των πλευρών ε, αυτής της Επιτροπής. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο αυτό το έγγραφο. Κύριε Γκρέχ, θυμάμαι τη συζήτηση που είχαμε στο Στρασβούργο όταν είχατε ξεκινήσει την έκθεση αυτή και πρέπει να πω ότι τα συμφραζόμενα αλλά και η φιλοσοφική και πολιτική προσέγγιση της εκθέσεώς σας θα βοηθήσουν πολύ την εργασία που κάνω ε, και ε, είχα, μπόρεσα να εμπνευστώ από τις προηγούμενες ε, επαφές και από την επαφή μαζί σας πολλά στοιχεία τα οποία θα ενσωματώσω στην έκθεσή μας και ευχαριστώ για τη συνεργασία. Θέλω να κάνω ορισμένα σχόλια για την έκθεση του Λουί Γκρέκ, διότι την έχω διαβάσει και χωρίς να σας απογοητεύσω κύριε Πρόεδρε σας και το ακροατήριό σας με λίγα λόγια θα σας πω πώς σκοπεύω να αναβαθμίσω τη δικιά μου έκθεση. Η έκθεση Γκρέχ κατά τη γνώμη μου έχει το μεγάλο προσόν να επιλέγει την ολιστική προσέγγιση για την ενιαία αγορά, πράγμα που είναι κάτι νέο για κοινοβουλευτικά έγγραφα και ε, για το γραπτό κείμενο γενικώς. Δηλαδή παρόλο που στη διατύπωση στην έκθεση κινείστε μεταξύ εσωτερικής και ενιαίας νομίζω ότι η ενιαία αγορά δίνει ένα πιο σαφές μήνυμα ε, για τρεις λόγους, δύο που ανέφερα ήδη το Δεκέμβριο και ο τρίτος διότι αν μιλούμε σε πολίτες μίας χώρας μέλους για την ενιαία αγορά πολύ δικαιολογημένα θα, θα καταλάβουμε ότι αναφέρεστε στην εσωτερική αγορά αυτής της χώρας. Επίσης, ε, ε, εκτός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ε, πρέπει να υπάρχει μία προσέγγιση αυτών των δύο ενιών η οποία ακόμη και αν δεν ισχύει ουσιαστικά διότι οι εσωτερικές μας επιχειρήσεις αμφισβητούν την ενία αγορά γιατί θεωρούν ότι δεν είναι αρκετά ολοκληρωμένη και ότι υπάρχει μία προσέγγιση η οποία δεν υφίσταται και δεν θα έπρεπε να ε, ε, υφίσταται αλλά ο τρίτος λόγος είναι μία πρόκληση δηλαδή ε, όταν μιλάμε για ενιαία στην αγορά προβάλλουμε μία πρόκληση πολιτική διότι όλοι έχετε ε, τονίσει τη δυσκολία να διεκπαιρεώσει κανείς αυτή, αυτό το δύσκολο έργο την ενιαία αγορά που δεν είναι στόχος, που είναι εργαλείο και συμφωνώ πλήρως και επιπλέον είναι πολύ διαφοροποιημένο και διάχυτο στοιχείο είχα τρομάξει όταν ανέλαβα σαν Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς ε, πρόκειτο για ένα εγκυκλοπαιδικό χαρτοφυλάκιο πολυσχηδές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βλέπουμε ότι είναι μια διάχυτη έννοια ε, η οποία όμως είναι δύσκολο να οδηγήσει σε συνοχή. Πρόκειται για μια ολιστική προσέγγιση και πιστεύω ότι η έκθεση Γκρέκ ε, ανταποκρίθηκε πάρα πολύ σωστά ε, σε αυτή την πρόκληση. Ε, όπως άλλωστε είπατε κύριε Πρόεδρε, ε, αν θέλετε να υπάρξει κάποια δράση, δεν χρειάζεται μόνο νομοθεσία για την ενιαία αγορά, αλλά θα χρειαστεί μία πράξη, ε, act ή action Μία πράξη λοιπόν ε, ε, νομοθετική ενδεχομένως ε, ή που να συγκεράζει και τα δύο στοιχεία για να προχωρήσουμε. Ποια είναι λοιπόν τα στοιχεία της ολιστικής προσέγγισης για την ενιαία αργορά που δεν έχουν αναπτυχθεί επαρκώς στην έκθεση Γκρέχ. Προσπάθησα να διαβάσω το κείμενο από αυτή την κριτική οπτική γωνία και πιστεύω ότι ορισμένα θέματα δεν έχουν αναπτυχθεί όσο θα μπορούσαν. Αλλά αυτό οφείλεται στο ε, το περιορισμό των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής ε, Εσωτερικής Αγοράς. Ε, διότι αυτό τονίζει όπως και εις την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι πρέπει να συγκεράσουμε τις δραστηριότητες των 14 γενικών διευθύνσεων που ασχολούν ασχολούνται με την ενιαία αγορά και στο Κοινοβούλιο χρειάζεται να αναλυθεί μια πιο ολιστική αντιμετώπιση για να ενισχυθεί ε, η προσπάθεια και βλέπουμε ότι αναφέρεστε εις ε, τις οδηγίες και τους κανονισμούς που αναφέρονται στην εσωτερική αγορά ε, και αναφέρεστε εις τους στα συμπληρωματικά στοιχεία αλλά και στα αντιφατικά στοιχεία τα οποία υπάρχουν. Υπάρχει μία διάσταση κοινωνική, ε, πολιτική, οικονομική, βιομηχανική ε, και μία εξωτερική η οποία γίνεται ε, όλο και πιο σημαντική διάσταση και που δεν άπτεται των δραστηριοτήτων της ε, δικιάς σας ε, επιτροπής αλλά ε, εγώ στη θέση σας δεν θα δίσταζα να προχωρήσω περισσότερο και να αναφέρω ότι και αυτά τα στοιχεία πρέπει να περιληφθούν για να καλύψουν όλη την ολιστική προσέγγιση. Όσον αφορά την βιομηχανική και την εξωτερική διάσταση θα κάνω ένα ακόμη σχόλιο συμφωνώ ότι ε, είναι σωστή ο προσανατολισμός εκθέσεως ΚΡΕΚ προς τον καταναλωτή κάθετος πολίτη και ε, λέει ότι πρέπει να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη ε, των ε, καταναλωτών και να επανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών που αισθάνονται ότι η ενιαία αγορά δεν έχει καλύψει και τα μη οικονομικά δικαιώματά τους και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις διότι βλέπετε όλο και περισσότερο ότι και επιχειρήσεις ακόμη και μεγάλες επιχειρήσεις είναι είναι πολύ σκεπτικοί ε, ε, αφιζητούν πάρα πολύ τις αρχές της ενιαίας αγοράς του παρελθόντος πράγμα το οποίο οφείλεται ή στη βιομηχανική και εξωτερική διάσταση διότι μεγάλοι πρόεδροι εταιριών ή στην Ευρώπη θα σας πούν ότι δεν έχουν, έχουν μεν πιστεί ότι η ενιαία αγορά είναι ένα σημαντικό εγχείρημα αλλά ε, πώς θα συνδυαστούν οι διάφορες πολιτικές με την ανάγκη του να έχει κανείς ε, ε, πανευρωπαϊκούς πρωταθλητές και πώς θα γίνουν αυτά σε ένα κόσμο όπου εφαρμόζονται αυστηροί κανόνες για την ε, ε, κρατική ενίσχυση ενώ οι κανόνες αυτοί δεν ισχύουν εκτός Ευρώπης. Υπάρχουν λοιπόν ε, σημαντικές αλλαγές οι οποίες πρέπει να γίνουν αλλά πάνω απ' όλα μία παιδαγωγική προσπάθεια για να εξηγήσουμε ότι δεν είναι αδύνατον να υπάρξουν ευρωπαϊκοί πρωταθλητές μέσα στα πλαίσια αυτών των κανόνων ότι η Ευρώπη πρέπει να αυξήσει τις προσπάθειές για να εφαρμόσει τις αρχές που διέπουν τις σχέσεις μεταξύ ε, των ε, κυβερνήσεων και των ε, πολιτών διότι του χρόνου θα έχουμε στη Γαλλία την προεδρία του GE όπου θα δοθεί η δυνατότητα να προβληθούν τα θέματα αυτά στη συνάντηση των G20 όπου ε, θα δούμε ότι οι χρηματοοικονομικές σχέσεις πρέπει να τονίζονται όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και γενικότερα. Και ε, τελειώνοντας και αναφέροντας λίγο τα στοιχεία της εκθέσεώς μου η προθεσμία για την υποβολή στον πρόεδρο Μπαρόζο είναι τέλη Απριλίου, δηλαδή πλησιάζομαι πολύ. Και όσον αφορά ε, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορώ ε, σε αυτή τη φάση να υπησέλθω σε λεπτομέρειες και να ε, προαναγγείλω τι συστάσεις ε, θα διατυπώσω. Θα έχω διάφορες συστάσεις να διατυπώσω, αλλά τα μέλη της Επιτροπής ΙΜΚΟ δεν θα εκπλαγούν όταν θα δημοσιευθεί αυτή η έκθεση για την ενιαία αγορά, διότι πιστεύω ότι έχετε μία πνεύμα πραγματική συνέργεια και ε, ε, ε, προσέγγιση στο θέμα αυτό και έχω εμπνευστεί πολύ από τα θέματα τα οποία έχουμε συζητήσει και άλλωστε στη συζήτηση που έχουμε σήμερα θα αντικατοπτρίζεται στην έκθεση αυτή. Διότι από την προηγούμενη συνάντησή μου ο προέβην σε πολλές διαβουλεύσεις όπως μου το ζήτησε ο πρόεδρος Μπαρόζο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πέραν της Επιτροπής ΣΥΜΚΟ που ήταν η Επιτροπή Κλειδί ε, με την ε, Επιτροπή Κρίσεως με ε, την Επιτροπή που οργανώνει το διάλογο με τα Εθνικά Κοινοβούλια και είχα συζητήσεις και με πέντε πολιτικές ομάδες ΕΛΚ, Σοσιαλιστές, Φιλελεύθεροι, Ευρωπαίους Συντηρητικούς και θα έχω ακόμη και και με την ΚΟΕ που δεν συνάντησα ακόμη. Ε, επίσης συναντήθηκα με τον πρόεδρό σας, τον κύριο Μπούζε και στα πλαίσια του Συμβουλίου Είχα ήδη ε, δύο συναντήσεις με τον πρόεδρο Βαν Ρομπόη ε, και ε, ανταλλαγές απόψεως με την Επιτροπή Εκοφήν και Ανταγωνιστικότητος και σε επίπεδο κρατών μελών με όλα τα κράτη-μέλη εντός των πλαισίων των συμβουλίων και με τους περισσότερους διμερός κατόπιν πρωτοβουλίες μου με τους υπουργούς τους που ε, συμμετέχουν στα Συμβούλια Εκοφήν και Ανταγωνιστικότητας και ε, βεβαίως με όλων των ειδών τους ενδιαφερόμενους πολίτες. Ε, λοιπόν, ε, από όταν συναντηθήκαμε τον Δεκέμβριο υπήρξαν δύο βασικά θέματα τα οποία προέκυψαν στη συζήτηση που αύξησαν την σημασία και έδωσαν μια νέα διάσταση στην ενιαία αγορά. Το ένα, κύριε Ράπτη, είναι η ελληνική κρίση. Η ελληνική κρίση αναφέρεται εις ε, ε, τα δημοσιονομικά θέματα της Ευρωζώνης αλλά είναι μία σαφής εκδήλωση ενό πιο βαθιού και πιο ευρέως προβλήματος που είναι η έλλειψη ε, παρκώς σοβαρής εκτιμήσεως της ενιαίας αγοράς αντιλαμβανόμαστε όλο και περισσότερα ότι η Ελλάδα έχει ένα θέμα ανταγωνιστικότητος το οποίο υποθάλπει και τα δημοσιονομικ... τις δημοσιονομικές της δυνατότητες και τις δυνατότητες χρηματοδοτήσεως, αλλά υπάρχουν στον πίνακα βαθμολόγησης ε, ε, και συμμορφώσεως ε, στοιχεία που δείχνουν ότι η Ελλάδα δεν πάει καλά όσον αφορά την ενσωμάτωση της οικονομίας της στην ενιαία αγορά. Δεν έχει λοιπόν επιτρέψει στην οικονομική ολοκλήρωση που που, που προσφέρει η ενιαία αγορά ε, να δυνατότητα να βελτιώσει την οικονομία της όπως έκαναν άλλα κράτη. Ε, αν υπάρχει επαρκής ανταγωνιστικό αναγωνισμός και ανοιχτή αγορά μπορεί κανείς να προχωρήσει καλύτερα. Και ένα άλλο στοιχείο το οποίο έχει προκύψει από την τελευταία συνάντησή μας είναι η οικονομική διακυβέρνηση κατόπιν της δραματικής ελληνικής κρίσης. Εάν λοιπόν αντιληφθούμε ότι και οι κρίσεις και οι δυσκολίες οι οποίες υπάρχουν στο δημοσιονομικό τομέα ή το νομισματικό τομέα βασίζονται ουσιαστικά σε ανεπαρκή ε, υποθάλπουσα στήριξη του ανταγωνισμού των αγορών τότε αντιλαμβάνεστε ότι και άλλωστε ο πρόεδρος Βαροπόη νομίζω ακολουθεί το ίδιο σκεπτικό ε, αντιλαμβάνεστε ότι το πρώτο στοιχείο για το Συμβούλιο και το πρώτο θέμα ε, για την ε, οικονομική διακυβέρνηση ε, είναι ο στόχος της οικονομικής εντάξεως ή στην ενιαία αγορά και αυτό όχι μόνο για την Ευρωζώνη παρόλο που είναι ιδιαίτερα σημαντικό όπως απέδειξε η ελληνική κρίση και όχι μόνον ότι ιδιαίτερος ή την Ευρωζώνη πρέπει να υπάρχει πλήρη στήριξη ε, και συμμόρφωση με την ενιαία αγορά για να μπορέσει κανείς να υποφεληθεί. Αυτά λοιπόν είναι λίγα σχόλια σχετικά με το πώς ε, θα παρουσιάσω ε, το σκεπτικό αυτό το οποίο νομίζω ότι είναι κοινό μεταξύ της Επιτροπής σας και μου και ε, πόσο από την τελευταία φορά που συναντηθήκαμε ε, αξιολογώ το θέμα της ενιαίας αγοράς το οποίο η σημασία αυξήθηκε πάρα πολύ και δεν είναι πλέον περιθωριοποιημένη. Θα ήθελα τέλος να τονίσω ότι όλοι θα πρέπει να είμαστε ευγνώμονες, εγώ τουλάχιστον είμαι, προς τον κύριο Γκρέχ που κατάρτισε αυτή την έκθεση που προσφέρει συγκεκριμένα στοιχεία και πρωτοβουλίες και είναι ε, ένα πολύ καλό μέσο μεταφοράς και εφαρμογής αυτής της ολιστικής προσεγγίσεως. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τον καθηγητή Μόντι για αυτή την στοχαστική και σε βάθος ανάλυση θα έλεγα κάποιον από τα θέματα που συζητήσαμε για αυτά σήμερα. Και αναμένουμε στο να δούμε την έκθεσή σας με συγκεκριμένες σαφείς συστάσεις για αυτά τα οποία για λόγους που γνωρίζουμε και κατανοούμε δεν έχουν ακόμα υποβληθεί αλλά θα υποβληθούν και θα μπορούσα να ζητήσω να σχολιάσετε ίσως πρώτου ξαναρχίσει η συζήτηση και πάλι. Φαντάζομαι ότι θα υποβάλλετε τα αποτελέσματα της έκθεσής σας <clears throat> στη σύνοδο του Ιουνίου σε σχέση με τα όσα είχε υπόψη ο κύριος Φαν Αλλά ξέρουμε ότι υπάρχει και ένα Συμβούλιο Ανταγωνισμού τέλη Μαΐου επίσης που προβλέπεται να διεξαρθεί τότε. Το ζητώ αυτό εξειδικευμένα επειδή τα χρειαζόμαστε για να τα εξετάσουμε σε σχέση με την τελική ψηφοφορία για την έκθεση Λουί Γκρέκ δίνοντας χρόνο στους συναδέλφους να υποβάλουν και από πλευρά τους ενδιαφέρουσες τροπολογίες, αλλά να μην καθυστερήσουμε βέβαια και με την ψηφοφορία, ώστε να υπάρχει χρόνος να ληφθούν υπόψη οι προτάσεις σε αυτή τη συζήτηση. Δεν γνωρίζω ακριβώ ποιε είναι οι δικέ σα προσδοκίε ε, για την δική σα ε, παρουσίαση και από πλευρά χρονοδιαγράμματό σα, αλλά θα θέλαμε να ευθυγραμμίσουμε τη δική μα δράση με αυτό το σκέλο ε, των δικών σα συστάσεων, ώστε να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε. Κύριο Μόντι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι προ το γενικό συμφέρον αυτό να προσπαθήσουμε να καταφέρουμε να επιτύχουμε να υπάρχει αυτή η σύμπτωση και ευθυγραμμισμός χρονοδιαγραμμάτων μεταξύ μας. Όσον αφορά εμένα τον ίδιο τώρα, η χρήση του δικού μου προϊόντος θα είναι στην διακριτική ευχέρεια φυσικά του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, στη συνέχεια. Εγώ θα υποβάλω σε αυτόν την έκθεση κατά τα τέλη Απριλίου. Ο ίδιος ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα αποφασίσει τι θα απογίνει στη συνέχεια και επί της ουσίας και υπό τους όρους των διεργασιών ή των διαδικασιών. Μπορεί να έχετε δει ίσως ότι στο πρόγραμμα εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που πολύ πρόσφατα υιοθετήθηκε υπάρχει μια ένδειξη υπάρχει μια αναφορά της Επιτροπής. Δεν, δεν θυμάμαι ποιος όρος χρησιμοποιήθηκε. Πρωτοβουλία νομίζω ή έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, που προβλέπεται ε, κατά τη διάρκεια του μηνός Μαΐου για να αν υπάρξει ανταπόκριση και συνέχεια στην έκθεσή μου από πλευράς της. Μπορεί κανείς να το φανταστεί, αλλά ότι θα γίνει αυτό, αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι είναι απόλυτα στη διακριτική ευχέρεια του Προέδρου Μπαρόζο. Μπορεί κανείς βέβαια να φανταστεί ότι μπορεί να περάσουν κάποια από αυτά στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου. Φυσικά ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου έχει εκφράσει μεγάλο ενδιαφέρον για αυτό το θέμα και μια και αναφερθήκατε στο Συμβούλιο Υπουργών Ανταγωνισμού από τότε που είχα συμμετάσχει την 1η Μαρτίου με, για ανταλλαγή απόψεων με τους ε, υπουργούς η Ισπανική Προεδρία του Συμβουλίου Υπουργών Ανταγωνισμού, Ανταγωνιστικότητας ανέφερε την πρόθεσή της να με προσκαλέσει τον Μάιο, νομίζω τέλη Μαΐου, κατά τη διάρκεια της σύγκλησης της Συνόδου των Υπουργών ε, για τον ανταγωνισμό σε σχέση με την ανταγωνιστικότητα όταν θα έχει υποβληθεί η έκθεση. Λυπούμε που δεν μπορώ να εξειδικεύσω περισσότερο και να είμαι πιο συγκεκριμένος επ' αυτού. Αλλά προφανώς ε, τώρα εμπλέκομαι ακριβώς σε μεγάλο βάθος στην εκπόνηση, στην σύνταξη της έκθεσής μου και όχι στην εμπορία, στην ε, προώθηση του τελικού μου προϊόντος. Ήταν όμως χρήσιμα αυτά που μας είπατε, λέει ο Πρόεδρος. Εντάξει, συνάδελφε, ας ε, ξαναρχίσουμε τη συζήτηση. Τώρα από πλευρά ε, των παρεμβάσεων. Νομίζω ότι ίσως θα μπορούσαμε να ολοκληρώσουμε τον πρώτο γύρο παρεμβάσεων με τους ευρωβουλευτές. Έχουμε μια μισή ώρα ακόμα και πολύ χρόνο και Επιτρέψτε μου να σας πω ποιοι είναι εγγεγραμμένοι. Και μετά έχω ένα δεύτερο γύρο παρεμβάσει Κυρία Ράπτη και κυρία Γκέπχαρτ. Νομίζω στον πρώτο γύρο θα περάσετε εσείς και ο κύριος Ροσφόρ στον δεύτερο γύρο και η κυρία Καράτσα στον πρώτο γύρο. Εντάξει, ξεκινάμε λοιπόν με τον καθηγητή Κορέντε Κάμπος παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Φυσικά θα απευθυνθώ περισσότερο στην έκθεση Λουίς Γκρέκ παρότι αν μου επιτρέπετε θα έχω ιδιαίτερη ευχαρίστηση να κάνω και κάποια αναφορά στην ε, εισήγηση, στην παρέμβαση του καθηγητού Μάριο Μόντι, που η παρουσία του σήμερα είναι κάτι για το οποίο εκφράζω την ικανοποίησή μου και ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω ότι η έκθεση Λουίς Κρέκ είναι μια σημαντική έκθεση και βρισκόμαστε σε σύμπτωση ευθυγραμμισμένη στις απόψεις ε, με τον τρόπο με τον οποίο προσέγγισε το πρόβλημα <clears throat> για τις προτεραιότητες, τον κέριο ρόλο που πρέπει να έχουν οι καταναλωτές. Φυσικά όλοι μας θα θέλαμε αυτή η έκθεση να είχε <clears throat> αναφορές ε, στο διεθνές εμπόριο, στα θέματα ανταγωνιστικότητας, ε, στα θέματα χρηματικών, χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Όλοι θα θέλαμε βέβαια να υπάρχει να υπάρχουν δύο λόγια, μια αναφορά για αυτά τα θέματα. Όμως, από την άλλη πλευρά, αληθεύει ότι αυτά για να γίνουν με προτεραιότητα θα έπαιρναν πολύ, πολύ χώρο που ε, δεν είναι ακριβώς τα θέματα τα οικονομικά ε, ή τα θέματα της έκθεσης. Γι' αυτό πρέπει να αποφύγουμε το σύνδρομο του ευχολογίου, του χριστουγεννιάτικου δέντρου με επιθυμίες και ευχές, όπου όλες οι ευχές και οι επιθυμίες μας θα θέλαμε να λυθούν υπόψη ως ευχολόγιο. Λοιπόν, είναι προφανές του λεχθέντος, ότι όλοι συμφωνούμε με τον κέριο ρόλο που έχει η αγορά ως μέσο, ως εργαλείο για την ικανοποίηση ατομικών της εξέλιξη των ατόμων και και της κοινωνίας συλλογικά. Και όχι να βλέπουμε την αγορά ως ένα αυτοσκοπό, τελικό αυτοσκοπό των κοινωνιών μας. Και η έκθεση σε αντίθεση με τα όσα έχουν αναφερθεί μέχρι τώρα, είναι πολύ περισσότερο από μια καλή βάση εργασίας. Είναι, θα έλεγα ακόμα, μια έκθεση που πρέπει και μπορεί να διαδραματίσει ένα κέριο ρόλο, όχι μόνο λόγω της ουσίας της, αλλά λόγω του παράλληλου χαρακτήρα της σύμπτωσης ε, των χρονικών συγκυριών σε σχέση με την έκθεση ακριβώς των θεμάτων του κυρίου Μόντι. Ο εισηγητής εφιστά την προσοχή για το κέριο θέμα θεμελιώδους σημασίας, ε, δηλαδή <clears throat> το κύριο εμπόδιο ή τον κύριο λόγο παρεμπόδισης ε, που είναι στα κράτη-μέλη, θεωρεί ο εισηγητής. Συμφωνώ εγώ με αυτό. Πιστεύω ότι τα κράτη-μέλη δεν είναι αρκετά ευαίσθητα. Δεν υπάρχει ακόμα μια ownership, ας το πω έτσι, μια κοινοκτημοσύνη, ένα κοινό όραμα για αυτή την ενιαία εσωτερική αγορά. Και ίσως αξίζει τον λόγο να ε, σκεφτούμε λίγο γιατί συμβαίνει αυτό. Κυρίως όταν τα κράτη-μέλη σε κάποια χρονική συγκυρία είδαν να φτάνει στις ε, Βρυξέλλες μια εισβολή, μια υποχρέωση ανοίγματο των αγορών, των διεθνών αγορών και των εσωτερικών αγορών, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών αγορών και υπηρεσιών, όπου θα λέγαμε ότι είναι περισσότερο γνωστές οι ε, ελλείψεις των αγορών, ε, τα ευάλωτα στοιχεία, για παράδειγμα κοινωνικές υπηρεσίες σε σχέση με την αργή βραδία πρόοδο εισάγοντας κάθε φορά όλο και περισσότερο εκείνα τα αγαθά και τις υπηρεσίες ε, διασυνοριακά όπου υπάρχουν λιγότερες ρήξεις, ρήγματα ή ελλείψεις στις αγορές θα καταλήγαμε σε κάποια ας το πω σχετική όχι απόρριψη αλλά θα καταλήγαμε σε αυτή την επιφύλαξη ή στον σκεπτικισμό που αντιμετωπίζουν την εσωτερική αγορά ε, σε σχέση ε, με την πρόοδο χώρε χώρες μας. Και γι' αυτό, αυτό το, αυτά τα βήματα έχουν πολύ μεγάλη σημασία και πρέπει να γίνουν. Ουσιαστικά σε σχέση με τον κύριο Μάριο Μόντι όταν είπε ότι οι, ε, ε, οι αγορές ε, είναι ένα σύνολο ένα συνονθήλευμα διαφορετικών και ετερόκλητων στοιχείων και διαφορετικών μεταξύ τους. Πρέπει να είμαστε λοιπόν επιλεκτικοί, να επιλέξουμε εκείνα τα στοιχεία που μπορούν να οικοδομήσουν πιο γοργά την ενιαία εσωτερική αγορά για να μην καταλήξουμε σε δυσφορία και απογοήτευση όταν βλέπουμε τον κατάλογο των χωρών και εκείνες τις χώρες που είναι πιο καθυστερικές καθυστερημένες στην υλοποίηση των οδηγιών στο εθνικό επίπεδο ή σε σχέση με θέματα ε, διεθνούς εμπορίου. Παράδειγμα, το ηλεκτρονικό εμπόριο, όπου είναι ένας τομέας όπου η θεωρία των μικρών βημάτων μπορεί να είναι ε, σημαντική. Και έχοντας ακριβώς το θέμα για την έκθεση του ηλεκτρονικού εμπορίου είχαμε και ένα workshop με τους εκπροσώπους ε, των τομέων και αυτό που είδαμε να διαπιστώνεται από αυτές τις επιχειρήσεις είναι ότι παρόλες ε, τις ε, διαφορές και αντιθέσεις παρόλες τις παρεκκλήσεις όσον αφορά το ΦΠΑ στις διάφορες χώρες ή την τον υποχρεωτικό χαρακτήρα να υπάρχει η καταχώρηση σε σχέση με το ΦΠΑ σε, διάφορε... σε διαφορετικές χώρες και σε σχέση με την, ε, το θέμα της ε, μη επαρκούς εμπιστοσύνη σε σχέση με τον τραπεζικό τομέα συνεχίζει να προχωρεί το ε, ηλεκτρονικό εμπόριο με διψήφιο κιόλας ποσοστό και συνεχίζει εδώ να προχωρά θα έλεγα βήμα προς βήμα και με ένα πιο ήρεμο χαρακτήρα βλέποντας αυτά τα μικρά βήματα υπερβαίνοντας και ξεπερνώντας τα προσκόμματα που μας οδηγούν σε παράλυση και με ένα πραγματικό πραγματιστικό τρόπο βρίσκοντας λύσεις. Στο τέλος τέλος θα ήθελα να απευθυνθώ στον Μάκομ Χάμπορ και να πω ότι πραγματικά εντυπωσιάστηκα Μάκομ με τον ενθουσιασμό που σας ε, εμπνέει σε σχέση με τον πρωταγωνιστικό ρόλο που πρέπει να ε, δοθεί σε σχέση με την ε, διάσταση της εσωτερικής αγοράς και την αναζωγόνησή της. Αυτό που μας προτείνει ο Λουί Γκρέκ σε σχέση με την μέθοδο σε τέσσερις φάσεις, σε τέσσερις άξονες βασιζόμενα ενδεχομένως στην ε, νομοθετική δράση ή και με διαφορετικό τρόπο γιατί είμαστε ένα ε, όργανο που το κύριο όργανο μας είναι η ε, δράση μας όσον αφορά την δραστηριοποίηση σε νομικό πλαίσιο. Δεν έχω την αναγκαία πείρα να γνωρίζω αν η ε, ένα νομοθέτημα όπως ε, η Single Market Act, το νομοθέτημα για την εσωτερική αγορά είναι το μόνο. Μου φαίνεται ότι δεν είναι ε, εδώ μόνο ένα μέσο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να δούμε την δυνατότητα παραλληλισμού ώστε να έχουμε πρωταγωνιστικό ρόλο για το Συμβούλιο για την Ενιαία Εσωτερική Αγορά ώστε να είναι οι προσπάθειές μας προς τον κοινό στόχο. Ευχαριστώ. Uh, σας ευχαριστώ πολύ. Και μια αναλογία έκανα σε σχέση με το νομοθέτημα αυτό μεταξύ νομοθετικών και μη νομοθετικών μέτρων. Δεν ήταν αναγκαστικά επικεντρωμένη στην νομοθετική δράση αυτή η παρατήρηση. Και θα το ξαναδούμε το θέμα με τις τροπολογίες επί του, της έκθεσης του κυρίου Γκρέκο. Κύριος Τριανταφυλλίδης. Κύριος Τριανταφυλλίδης μετά Κρόισμαν Τόρμερ και έτσι ολοκληρώνουμε τον πρώτο γύρο. Και στο δεύτερο γύρο Γκέπχαρτ και κυρία Ράπτη, Και νομίζω ότι θα πρέπει πιθανότατα και προφανώς ο κύριος Γκρέκ θα επανέλθει στο τέλος ε, των, γύρων αυτών στη συζήτηση και μετά αν θα θέλει η κυρία Βάμπταμ να συμβάλλει στη συζήτηση και να λάβει τον λόγο αν επιθυμεί ο κύριος Μάριο Μόντι για τελικά σχόλια αν έχει. Σα ευχαριστώ Πρόεδρε. Φυσικά ζήτησα τον λόγο για να αντιδράσω στην έκθεση Γκρέκα, έχοντα ε, το νόημιο να ακούσω τι παρατηρήσει του ε, καθηγητή Μότι θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για τα σχόλια που έκανε και όσον αφορά την έκθεση του κυρίου Γκρέκ αλλά και την δική του έκθεση. Δεν έχω καμιά αμφιβολία. Θα έχουμε μια συνάντηση μαζί του, η δική μου κοινοβουλευτική ομάδα μαζί του. Ήδη έχουμε αποστείλει μια επιστολή προ αυτόν με κάποιες απόψεις ε, όσον αφορά τις θέσεις μας ε, για το δικό του εγχείρημα. Αλλά προσβλέπουμε επίσης και σε διμερείς ε, συζητήσεις και επαφές που θα ακολουθήσουν. Θα ήθελα τώρα πρώτα απ' όλα να τονίσω το σχόλιο το οποίο έκανε ότι υιοθετεί και ενστερνίζεται την φιλοσοφική προσέγγιση της έκθεσης του Λουίγκρεκ διότι καθελκύοντα εκ νέου, αναζωογονώντα την ε, ενιαία εσωτερική αγορά, με ιδιαίτερη χαρά βλέπουμε ότι αυτό θα γίνει. Γίνεται με ένα νέο τρόπο νοοτροπία και προσέγγιση. Και ο κύριο Γκρέκ ουσιαστικά ενέταξε στην έκθεσή του αυτά που πιστεύουμε και εμεί ε, ω αρχέ. Και πρέπει εδώ να τονίσω ότι οι ε, φιλόσοφοι, οι διανοούμενοι τη αριστερά ήταν πραγματικά πάρα πολύ σκεπτικιστέ και επιφυλακτικοί όσον αφορά την ενιαία εσωτερική αγορά ω σύνολο. Χαιρόμαστε τώρα ότι υπάρχει ένα νέο όραμα, μια νέα πολιτική προσέγγιση στην ανακαθέλκυση της εσωτερικής αγοράς. Φυσικά θέλω να τονίσω το γεγονός ότι με ιδιαίτερη ικανοποίηση το βλέπω ότι η έκθεση του κυρίου Γκρέκ θέτει στο επίκεντρο το, αυτού του νέου οράματο του καταναλωτές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσει. Και επίση εμπλέκει του πολίτε γενικά σε αυτό την προσέγγιση σφαιρικά. Είναι σημαντικό να μην σταματάμε, να μην αυτό το οποίο ε, έχει, είναι συμφέρον των επιχειρήσεων, των χρηματοοικονομικών κύκλων, αλλά να γίνεται λόγος για την προστασία των ε, καταναλωτών και των δικαιωμάτων των πολιτών. Και ολοκληρώνω αναφέροντας ότι είναι ιδιαίτερη ευχαρίστηση για μας να βλέπουμε ότι σε αυτή τη νέα πολιτική προσέγγιση θέτει την κοινωνική ενιαία εσωτερική αγορά ως στο επίκεντρο, ως σημαντικό υπόβαθρο και ότι οι πολίτες έτσι, οι καταναλωτές μπορούν να διαδραματίσουν, θα διαδραματίσουν για την εσωτερική αγορά ένα μεγάλο, πολύ σημαντικό ρόλο. Θέλω να ευχαριστήσω και τους δύο, και τον κύριο Μόντι και τον κύριο Γκρακή αυτό. Ευχαριστώ. Uh, now, Mrs. Η κυρία Τούν παρακαλώ. Um, Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Σήμερα σε πολλές συζητήσεις και παρεμβάσεις ε, αναφέρθηκε πόσο σημαντικό είναι το στοιχείο Τη ενιαία εσωτερική αγορά. Πόσο σημαντική είναι η Ευρώπη σφαιρικά. Όμως διαπιστώνουμε επανειλημμένα ότι αυτό το μήνυμα δεν περνάει στου πολίτε, Πιο πριν είπε κάποιο ότι θα έπρεπε η Ευρώπη να περάσει στην καρδιά των πολιτών, να δώσουμε ένα πρόσωπο ευδιάκριτο στην Ευρώπη και διαπιστώνουμε επανειλημμένα αν πάρουμε τη Γερμανία 99 ευρωβουλευτέ και σχεδόν ε, ε, 100 εκατομμύρια πολίτε είναι αυτό ιδιαίτερα σημαντικό. Πρέπει να δώσουμε συνέχεια σε αυτή την πρόταση. Πρέπει να το καταφέρουμε το όφελος, τα θετικά στοιχεία της Ευρώπης, επιτόπου να τα περάσουμε στους πολίτες μας, ε, στις χώρες μας. Πρέπει να κάνουμε μια διαχείριση, ας το πω έτσι, με τέτοιο τρόπο ώστε οι τοπικές εφημερίδες να αναφέρουν τα ευρωπαϊκά ε, τεκτενόμενα. Διαπιστώνουμε ότι έχουν ε, απεσταλμένους, έχουν ανταποκριτές και εδώ είναι μεγάλες περιφερειακές εφημερίδες στις Βρυξέλλες παρούσες, όμως οι, πιο, οι ευρύτερες εφημερίδες σε τοπικό περιφερειακό επίπεδο είτε δεν αναφέρουν καν τι γίνεται γίνεται στις Βρυξέλλες ή με αρνητικό τρόπο αναφέρονται στα όσα γίνονται εδώ. Πρέπει να είναι στη σύγχρονη εποχή η δυνατότητα να είναι δεδομένη να περνάμε αυτά τα θετικά στοιχεία στους ε, πολίτες. Παράδειγμα, τέλη περιαγωγής όσον αφορά την κινητή τηλεφωνία. Πολύ θετικό αυτό για τους πολίτες και πολύ θετική η ας το πω, παρουσίαση στους πολίτες. Καθώς επίσης και σε χρηματοοικονομικές συναλλαγές με τις τράπεζες, ανάληψη μετρητών για παράδειγμα ή εμβάσματα και αυτό να μπορεί να περάσει. Έχουμε εδώ και για παράδειγμα και την πρόταση να καθορίζεται ε, τον καθορισμό ε, τελών 5 ε, ευρώ και όταν συζητάτε αυτό επί τόπου περιφερειακά λέγεται υπάρχει κόστος όταν γίνονται αναλήψεις τότε το κόστος αυτό από ταμιευτήρια για παράδειγμα καλύπτεται αλλά υπάρχει ένα πολύ μεγάλο δίκτυο στη Γερμανία και δεν βλέπουμε να υπάρχει λόγος το κόστος ε, το οποίο δεν επομίζονται μεγάλε τράπεζε, να το επομίζονται οι πολίτε. Και πρέπει φυσικά να υπάρξει ρύθμιση διευθέτηση του κόστου. Είναι ένα θέμα που πρέπει οι τράπεζε οι ίδιε ε, να το ρυθμίσουν. Δεν έχει κανένα νόημα να επιβαρύνονται οι Ευρωπαίοι πολίτε με τέτοια τέλη. Και όταν στη Γερμανία για 5 ευρώ ανάληψη ε, υπάρχει τέτοια ρύθμιση, πώ είναι δυνατόν να μην υπάρχει μια ρύθμιση ευρωπαϊκή. Είναι θέμα τεχνική ρύθμιση. Ε, το θέμα της ρύθμισης των τελών. Δεν έχει νόημα τους Ευρωπαίους πολίτες να τους επιβαρύνουμε στο εξωτερικό με μεγαλύτερα τέλη. Με αυτό το παράδειγμα θέλω να δείξω ότι μπορούμε να δώσουμε ένα πρόσωπο στην Ευρώπη, ώστε στους πολίτες, στους καταναλωτές, όπως λέγεται, να υπάρχει σαφές το πλεονέκτημα, να τους δίνεται η εικόνα της Ευρώπης ως πλεονεκτήματος και πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για παράδειγμα αυτά τα πλεονεκτήματα στην ενιαία ζώνη, νομισματική στη ζώνη του ευρώ για παράδειγμα στο Βερολίνο, στη, σε αρμόδια ε, συνάντηση τελωνίων, εκφράστηκε το παράπονο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα, είναι πολύ λίγο γνωστά τα όσα γίνονται σε σχέση με τα τελωνιακά. Και αυτό είναι πάλι ένα θέμα της ε, επεξεργασίας και πράγματι η τελωνιακή αυτή υπηρεσία είναι πολύ λίγο γνωστή, έχει σχετικά λίγους συνεργάτες, όμως σε σχέση, και αυτό δείχνει η μελέτη, ε, έχει για παράδειγμα μεγάλο έργο για να ικανοποιούνται οι ανάγκες των πολιτών. Και με το, την οδηγία περιπαροχής ε, υπηρεσιών θα πρέπει να δούμε ότι θα υπάρχουν πολλά περισσότερα παράπονα τα οποία θα υποβάλλουν ενδιαφέρονται από τους πολίτες της Ευρώπης. Πρέπει να γίνει πιο γνωστή αυτή η ε, υπηρεσία. Πρέπει να περάσουμε και στα κρατήρια και στις περιφέρειες. Και αυτό πάλι είναι ένα σημείο όπου οι πολίτες αλλά και οι επιχειρήσεις μπορούν κυρίως να δουν ποια προτερήματα απορρέουν από την Ευρώπη συνολικά. Ολοκληρώνοντας θέλω να πω πρέπει να τα καταφέρουμε να δώσουμε μια εικόνα, ένα πρόσωπο σε αυτή την Ευρώπη. Αυτό δεν μπορούν μόνο οι εκπρόσωποι των κοινοβουλίων επιτούν, αλλά πρέπει να υπάρξει ένα καλύτερο marketing μια καλύτερη προώθηση, διαφήμιση, ώστε να μπορέσει να περάσει αυτή η εικόνα στον τοπικό τύπο και ε, τα δημοσιεύματα και να μπορούν να υπάρχουν δημοσιεύματα, για παράδειγμα κάθε εβδομάδα, κάθε δύο εβδομάδες, τι δίνει η Ευρώπη, τι προσφέρει η Ευρώπη στους πολίτες. Να, μπορούν, να, να μπορούμε να γνωρίζουμε ότι όταν πρόκειται για μια υπηρεσία marketing που θα λέει και θα ε, διαφημίζει ποια είναι τα προτερήματα της Ευρώπης χειροπιαστά, είμαι πεισμένος ότι θα περνούσε το μήνυμα στους πολίτες. Διαβάζονται πολύ περισσότερο αυτά τα έντυπα και θα δίναμε μια εικόνα στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Uh, thank you, Σας ευχαριστούμε. Η κυρία Τούν τώρα λοιπόν παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση βλέπω ότι χάρη στην έκθεση του κυρίου Γκρέκ έχουμε μια τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση σήμερα και χάρη επίσης και στον κύριο Μόντι τον ίδιο και ελπίζω ότι αυτό θα είναι μια, ε, ας ε, ένα θέμα το οποίο θα τύχει συνέχειας και αυτό επειδή όταν επαναλαμβάνουμε τον όρο δυσφορία ή δυσαρέσκεια όσον αφορά τους Ευρωπαίους πολίτες σε αυτή τη συζήτηση δημιουργείται κάποια θλίψη. Δημιουργείται θλίψη επειδή η ενιαία εσωτερική αγορά είναι, φαίνεται ότι είναι η μεγαλύτερη, ε, ε, το μεγαλύτερο επίτευγμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι κολοσσίων διαστάσεων επίτευγμα. Και όταν ακούμε ότι υπάρχει απογοήτευση από πλευρά των πολιτών, εγώ πιστεύω ότι είναι απογοητευμένοι οι Ευρωπαίοι πολίτε με την εσωτερική αγορά για δύο λόγου κυρίω. Πρώτον, επειδή οι πληροφορίε ήταν ανεπαρκεί για να κατανοήσουν το τι έγινε. Και κάποια φλέγοντα θέματα μπορούν να θεωρηθούν ως επιτυχίες, αλλά πολλοί πολίτες δεν ξέρουν πώς να υποφεληθούν από την ενιαία εσωτερική αγορά. Κάποιοι πολίτες έχουν ελιπός πληροφορηθεί και από την άλλη πλευρά η μεταφορά του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου δεν ήταν απόλυτα επιτυχής και πλήρης Σκέφτομαι λοιπόν και λέω, αν πραγματικά γνωρίζουμε πραγματικά πολλά για τις ελευθερίες, τις θεμελιώδεις ελευθερίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για παράδειγμα για την υγειονομική περίθαλψη, αναφέρθηκε αρκετές φορές σε αυτή τη συζήτηση το θέμα των υπηρεσιών υγείας. Για παράδειγμα, αν ασφαλιστικές εταιρείε θα είναι ανοιχτές και θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στην εσωτερική αγορά. Αν θεραπευτές και ε, νοσηλευτές θα μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Αν θα υπάρχει αμοιβαία αναγνώριση διπλωμάτων για παράδειγμα αν τα φάρμακα και τα σκευάσματα θα είναι ε, προσπελάσιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τους πολίτες. Αυτό θα πρόσθεται πρόσθετη αξία, προστιθέμενη αξία στην Ευρωπαϊκή Εσωτερική Αγορά. Επίσης και οι επιχειρήσεις θα ήταν σε καλύτερη θέση για να μπορούν να λειτουργούν αποτελεσματικά. Αυτές τις δύο πτυχές λοιπόν να τις λάβουμε υπόψη από κοινού. Και αν οι τράπεζες, τα τραπεζικά ε, ιδρύματα θα μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Αν μπορώ εγώ να κάνω την πληρωμή μου με την EC κάρτα, Εντάξει, πολύ καλά. Αλλά ως πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έπρεπε να έχω τουλάχιστον τρεις ε, πιστοτικές κάρτες, τραπεζικές πιστοτικές κάρτες. Διότι με μία και μόνο δεν, μπορώ, δεν μπορεί κανείς να δράσει πανευρωπαϊκά. Πρέπει λοιπόν να τα καταφέρουμε να δώσουμε στους πολίτες αυτά που χρειάζονται για να μην υπάρχει αυτή η δυσφορή, η δυσαρέσκεια. Έχουμε μεγάλη πορεία να διανύσουμε. Όταν βλέπω τη ζωή μου καθημερινά εδώ στις Βρυξέλλες, ας πάμε και ας δούμε τα προβλήματα χειροπιαστά. Υπάρχει διαφορά για παράδειγμα στην χρέωση των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων και σε σχέση και με την περιαγωγή. Ας κάνουμε λόγο για ανταγωνιστικότητα όπου θα διαγωνίζονται επιχειρήσεις και όχι κράτη-μέλη. Αν πάρει κανείς διαφορετικές χώρες, Βέλγιο και Πολωνία για παράδειγμα, οι τιμές, η χρέωση είναι πολύ διαφορετική. Εδώ λοιπόν είναι πολύ διαφορετικές. Δεν μπορεί να γίνεται λόγος λοιπόν για μια εσωτερική αγορά με κοινού όρου και ε, ε κοινέ προδιαγραφές και με την ε, δυνατότητα να έχω επαφή για παράδειγμα μέσω διαδικτύου τη, στην εταιρεία μου με ιδιαίτερη περηφάνεια λέω είμαι Ευρωπαία πολίτης όμως πολλές φορές υπάρχει εδώ και απογοήτευση κάνουμε λόγο για το ηλεκτρονικό εμπόριο λοιπόν αν θέλουμε να αγοράσουμε ένα εμπόρευμα, ένα προϊόν από μια διαφορετική χώρα παίρνουμε την πληροφορία ότι δεν βρίσκεται λέει προ, σε, σε πρόσβαση σε εσά αυτό το προϊόν γιατί δεν είναι στην περιφέρειά σας ποιες δυνατότητες υπάρχουν προσεγγίζουμε τις θερινές διακοπές και θα υπάρχει διαφορετική χρέωση όσον αφορά τις ε, πτήσεις ανάλογα με το που βρίσκεται κανείς και που έχει την έδρα του. Αν κάποιος βρίσκεται στο Λονδίνο πρέπει να αγοράσει το εισιτήριό του στο Λονδίνο ή στο Ηνωμένο Βασίλειο με πιστοτική κάρτα για παράδειγμα που έχει εκδοθεί στο ίδιο αυτό κράτος στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό το εισιτήριο δεν μπορεί να το αγοράσει κανείς ε, σε άλλη χώρα χρησιμοποιώντας άλλη προέλευση πιστοτική κάρτα από άλλο κράτο Υπάρχουν πάμπολοι λόγοι λοιπόν Λοιπόν, για τους οποίους η πορεία που πρέπει να διανύσουμε είναι μακρότατη. Πρέπει να συνεργαστούμε στενά με τα εθνικά κοινοβούλια και να δούμε πώς μπορεί η κοινοτική αυτή πορεία να ευοδοθεί. Ε, στόχος μας και ρόλος μας είναι να δημιουργηθεί η σωστή ατμόσφαιρα, ο σωστός περίγερος ή περιβάλλον, ώστε να εμπλακούν οι πολίτες και να μπορέσουμε να παράσχουμε στους πολίτες μας τις πληροφορίες για το πώς θα μπορούν Πόσοι θα έπρεπε και μπορεί να λειτουργήσει η εσωτερική αγορά. Δεν είναι απειλή η εσωτερική αγορά. Σίγουρα δεν δημιουργεί απειλέ στου Ευρωπαίου πολίτε. Είναι πιθανότατα μία από τι μεγαλύτερε ευκαιρίε για μα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Η κυρία και είναι και ο Κάρας εδώ είναι ο σκιώδης εισηγητής, οπότε θα τον βάλω στον πρώτο γύρο, μαζί και με την κυρία Ράπτη. Αλλά θέλουμε και λίγο χρόνο για να ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και τον κύριο Γκρέκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς να συγχαρώ το, να χαιρετήσω το όραμά σας για μια νέα πολιτική πρωτοβουλία προκειμένου να γίνουν πιο φιλικοί άνθρωποι για την εσωτερική αγορά. Και χαίρομαι που βλέπω τον κύριο Μόντι να συμφωνεί, αλλά και πολλούς από τους συναδέλφους γιατί νομίζω ότι πρέπει να βρούμε δημιουργικούς τρόπους για να το δείξουμε αυτό. Επίσης μου άρεσε και η εικόνα της κυρίας, αλλά σίγουρα αυτή η κυρία πρέπει να είναι και πολύ σκληρή και ισχυρή για να μπορέσει να ανταγωνιστεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Και αυτό είναι το βασικό, αυτό είναι το πρόβλημα της Ευρώπης. Πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί, δηλαδή ποιότητα, καινοτομία, τεχνολογία. Επίσης χάρηκα που άκουσα ότι ο κύριος Μόντι θεωρεί ότι πρέπει να υιοθετήσουμε ολιστική προσέγγιση. Κατά τη γνώμη μου αυτό πρέπει να το συμπεριλάβεις Λουίς στην έκθεσή σου. Στην εσωτερική μας συζήτηση αντιπαραθέτουμε την ανάπτυξη και την ευημερία. Σας υπενθυμίζω ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η ραχοκοκαλιά της εσωτερικής αγοράς. Είναι το φως στην άκρη του τούνελ. Είναι ο τρόπος για να επανέλθουν οι θέσεις εργασίας στην Ευρώπη πρέπει να βρούμε κοινωνικές πολιτικές. Καλό είναι να μιλάμε για την κοινωνική διάσταση της Ευρώπης, αλλά ποιος θα χρηματοδοτήσει την ευημερία. Χρειαζόμαστε οικονομική ανάπτυξη για να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε τις κοινωνικές πολιτικές. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε αυτή την ιδεολογική αντιπαράθεση μεταξύ ευημερία και ανάπτυξης. Επίσης πρέπει να συνεχίσουμε το άνοιγμα αντί για τον προστατευτισμό, μείωση της γραφειοκρατίας, εφαρμογή του Small Business Act και διευκόλυνση των επιχειρήσεων. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να ενσωματώσουμε και πολύ σωστά το δείξετε με το παράδειγμα της Ελλάδας. Το κόστος της μη εφαρμογής της ήδη εγκριθήσας νομοθεσίας και επίσης πρέπει να πιέσουμε τα κράτη-μέλη να είναι διαφανή στην εφαρμογή της υπάρχουσας νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά. Το όνειρό μου, αν όχι το όραμα, είναι ότι θα μπορέσουμε να δείξουμε στους πολίτες ότι η εσωτερική αγορά δεν είναι για τις επιχειρήσεις γιατί και εδώ έχουμε μια ιδεολογική αντιπαράθεση όπου κάποιοι θεωρούν ότι ό,τι είναι καλό για τις εταιρείες είναι κακό για τους πολίτες και το αντίστροφο. Αυτή την οτροπία πρέπει να την υπερβούμε. Πρέπει να δείξουμε ότι η εσωτερική αγορά μπορεί να είναι κατάσταση όπου κερδίζουν όλοι και οι εταιρείε και οι πολίτες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριο Κάρας. Πρόεδρε, Αγαπητέ κύριε Μόντι, θα ήθελα να πω ότι διαρκώς θα έπρεπε κανείς σε σχέση με τις συμβουλές σας για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για την εσωτερική αγορά θα έπρεπε να ε, χρησιμοποιεί τις ε, ιδέες σας. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Γκρακ για την καλή ε, συνεργασία, για την καλή δουλειά που έγινε. Αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να δημιουργήσουμε αιτήματα τα οποία θα θέτουμε προς τον εισηγητή, επειδή η έκθεση έχει δοθεί προς μετάφραση. Θα έπρεπε τα πράγματα τα οποία απομένουν και εκκρεμούν υπό το δικό μας πρίσμα με τροπολογίες να τα διατυπώσουμε ώστε να μπορέσουμε να δούμε τι μπορεί να γίνει σε σχέση με τα αιτήματα αυτά των τροπολογιών. Νομίζω αυτή είναι η σωστή διεργασία τώρα. Δεν είναι λοιπόν δική του, ας το πω έτσι, δεν εκκρεμεί κάτι από πλευρά του, έχει κάνει την πρότασή του. Εμείς πρέπει να δούμε τι μπορούμε τώρα να ε, συμπληρώσουμε. Με τον κύριο Μόντι, το πρόβλημα που έχω αυτή τη στιγμή είναι ότι πολύ σωστά συζητάμε μαζί σας για τις προτάσεις για την ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς και την υλοποίηση, την εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνας σε αυτή την εσωτερική αγορά, σε αυτή τη νέα προσπάθεια για την εσωτερική αγορά. Από την άλλη πλευρά έχουμε τη στρατηγική για την Ευρώπη 2020 και δεν έχω καθόλου αποκομίσει την εντύπωση μέχρι τώρα ότι μεταξύ της δικής σας ομάδας εργασίας και της στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020 στη συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Συμβούλιο και στην Ευρωβουλή υπάρχει διασύνδεση μεταξύ μας, μεταξύ των προτάσεων. Διότι αυτή η εσωτερική αγορά που έχει τόσο τεράστιο δυναμικό ακόμα είναι ένα πολύ σημαντικό μέσο, ένα εργαλείο για την υλοποίηση της στρατηγικής του 2020. Και σε σχέση με τη στρατηγική του 2020 για την Ευρώπη, αυτή δεν είναι ας το πω έτσι, ένας αυτός Είναι ένα μέσο, είναι ένα εργαλείο να αντιμετωπίσουμε την διεθνή χρηματοοικονομική κρίση και τον, την παγκοσμιοποίηση. Αυτή η συγκεκριμενοποίηση με χειροπιαστά προγράμματα και σχέδια, με αναγκαία ευρωπαϊκά μέσα που θα είναι συνεκτικά μεταξύ τους, αυτό λείπει αυτή τη στιγμή. Καθορίζουμε πολλούς στόχους, πολλές επιθυμίες. Το χρονοδιάγραμμα όμως για την υλοποίηση αυτών των σχεδίων πεδίων, των μέσων, των εργαλείων και η διασύνδεση μεταξύ τους λείπει. Είναι πολύ αποδυναμωμένο αυτό το στοιχείο. Δεύτερον, πιστεύω ότι πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ, μια και σε πολλούς τομείς που έχει ανάγκη να υπάρξουν η εσωτερική αγορά, δεν υπάρχει ακόμα ευρωπαϊκή αρμοδιότητα. Κοινωνικά θέματα, πολιτικά θέματα, θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, θέματα φορολογικά, δεν είναι ευρωπαϊκή αρμοδιότητα. Πολλά ζητάμε να γίνουν, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να τα επιτελέσουμε με δικές μας αρμοδιότητες. Χρειάζεται εδώ ηγετικός ρόλος, leadership της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω στις προτάσεις σας να προβλέπετε την εμπλοκή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως νομοθέτη, ως συνομοθέτη, ώστε ο αναγκαίος συντονισμός να διασφαλίζεται και να μην καταλήγουμε σε ένα νέο διακυβερνητικό πλαίσιο εκτός και παράλληλα με τα κοινοβούλια, διότι έτσι δεν θα πετύχουμε την Ευρωπαϊκή ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά των πολιτών. Και αυτό είναι το σημαντικό για μένα. Κοινοβούλιο και πολίτες να μπορέσουν να συγκλίνουν, να διασυνδεθούν με διασύνδεση που είναι αναγκαία. Και αυτό είναι το πρόβλημα που έχουμε με τα κράτη-μέλη. Ο πολίτης είναι πολύ πιο μακριά από ότι έχει πάει πολύ πιο πέρα από ότι πολλές κυβερνήσεις. Διότι για τις πρωτοβουλίες που λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα θέματα αρμοδιότητας ε, στα θέματα εσωτερικής αγοράς, πολλές φορές τα κράτη τα θεωρούν ανάμειξη στις εσωτερικές τους αρμοδιότητες, διότι δεν έχουν δημιουργηθεί τα αναγκαία υπόβαθρα ως βάση. Πρέπει να πούμε τα σίκα σίκα και τα σκάφη σκάφη και πρέπει να υπάρξει αυτή η αλληλοδιασύνδεση και η αλληλοσυνάρτηση. Σας ευχαριστώ για το ε, διανοητικό έργο που επιτελείτε, για τις ε, προτάσεις που εκπονείτε και πρέπει τις τέσσερις αυτές ελευθερίες και να έχουμε και την πέμπτη ελευθερία, την εκπαίδευση κατά κατάρτιση, επιστήμη, έρευνα και ανάπτυξη και καινοτομία ώστε αυτά να μπορέσουν να προαχθούν ως προτεραιότητες έναντι των πολιτών και να μπορέσει η Ευρώπη να αντιμετωπίσει τον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κάρας πριν έρθετε είχαμε συζητήσει πολύ το γεγονός ότι η Ευρώπη 2020 δεν επικεντρώνεται περισσότερο στο θέμα. Περνάμε στο δεύτερο κύριο και παρακαλώ αγαπητοί συνάδελφοι να είστε σχετικά σύντομοι γιατί θέλουμε να μπορέσει να απαντήσει και η Επιτροπή και να έχει και λίγο χρόνο ο κύριος Κρέχα για να συνοψίσει. Η κυρία Ράπτη πρώτα. Ευχαριστώ και πάλι κύριε Πρόεδρε. Τέσσερα σημεία πάρα πολύ σύντομα. Το πρώτο είναι το εξής. Προηγουμένως έκανα δύο ερωτήσεις στον καθηγητή κύριο Μόντι. Ε, πώς θα προσπαθήσει να μετατρέψει το δίλημα αγορά ή κοινωνία αλληλεγγύης σε ψευτοδίλημα. Και το δεύτερο, με ποιο τρόπο θα προσπαθήσει να ξανακερδίσει τον Ευρωπαίο πολίτη. Από την τοποθέτησή του νομίζω ότι πρέπει να αισιοδοξώ και θα περιμένω με αγωνία αλλά και με ελπίδα το τελικό κείμενο της έκθεσης. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι τον άκουσα να μας λέει ότι ήρθε σε επαφή με διάφορες επιτροπές και διάφορους ειδικού. Ε, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, αλλά νομίζω ότι δεν άκουσα στις επαφές που είχε να έχει συζητήσει με κοινωνικούς φορείς με κάποιον από την επιτροπή απασχόλησης με κάποιους από την επιτροπή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βάζω αυτή την πτυχή μέσα στον προβληματισμό γιατί είναι και αυτά ζητήματα που έχουν να κάνουν με το κοινωνικό πρόσωπο της ευρώπης. το τρίτο ζήτημα έχει να κάνει με την αναφορά του στην ελληνική κρίση ε, τον άκουσα με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και απλώς θέλω, αν μου επιτρέπετε, να σημειώσω ότι η ελληνική κρίση έχει μια ευρωπαϊκή διάσταση και να θυμίσω ότι χθες άκουσα με πολύ μεγάλη ικανοποίηση τον κύριο ρομπόι να λέει ότι από αυτή την υπόθεση της ελλάδας η ευρώπη διδάχτηκε και διδάχτηκε μεταξύ άλλων το να προλαμβάνει την πρόληψη. Γιατί θυμίζω ότι πάρα πολλά πράγματα συνέβαιναν κακώς στην Ελλάδα, αλλά η Επιτροπή έκανε ότι δεν έβλεπε. Ή δεν έβλεπε όντως, δεν ξέρω. Και τέταρτο και τελευταίο. θυμίζω καθηγητά ότι στην Ελλάδα έχουμε μια καινούρια κυβέρνηση σοσιαλιστική εδώ και μερικούς μήνες. Έχουμε μια κυβέρνηση που κάνει μια τεράστια προσπάθεια. Ε, πάρα πολύ σωστά σημειώσατε ότι έχουμε μια καθυστέρηση στο να ενσωματώσουμε το κοινοτικό δίκαιο, τις οδηγίες, στο εσωτερικό δίκαιο. Επειδή μέχρι το 2009 που ήρθα εδώ ήμουνα εθνική βουλευτής για πέντε χρόνια, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι μέσα στην Ελληνική Βουλή ε, το πασόκ ως αντιπολίτευση είχε εγκαλέσει πάρα πολλές φορές την κυβέρνηση για αυτή την καθυστέρηση και επειδή συνήθως λέμε ότι αυτά κάποια πράγματα τα λες όταν είσαι αντιπολίτευση αλλά τα ξεχνάς όταν γίνεσαι κυβέρνηση θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι αυτό δεν συμβαίνει. παράδειγμα τώρα τους επόμενους μήνες και σίγουρα νομίζω στον τον Ιούνιο, για παράδειγμα, η οδηγία για το άνοιγμα των επαγγελμάτων θα ενσωματωθεί με νομοθέτημα στο ελληνικό δίκαιο. Βάζω τελεία και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you very much. Και εμείς σας ευχαριστούμε για τις διαβεβαιώσεις. Κυρία Γκέπχαρτ. Ευχαριστώ. Είχα προηγουμένως τη δυνατότητα να μιλήσω για την έκθεση του Λουί Γκρέχ, αλλά τότε δεν είχε μιλήσει ο κύριος Μόντι και θα ήθελα και εγώ να αντιδράσω, γιατί είναι ε, ε, ένα βασικό στοιχείο για τη συζήτηση. Εχθές όμως στη συνεδρίαση των συντονιστών είπαμε ότι η έκθεση Λουί Γκρέχ θα είναι μία συμβολή μας για την στρατηγική του 2020 και έτσι πρέπει να προβληθεί διότι ε, δείχνουμε πως θέλουμε να διαμορφώσουμε την εσωτερική αγορά για τον καταναλωτή και τον πολίτη και γι' αυτό είναι πολύ σημαντική για τη συζήτηση την οποία διεξάγουμε αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν δύο θέματα που ανέφερε ο κύριος Μόντι και θέλω να σχολιάσω. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας όταν λέτε ότι η οικονομική κρίση απέδειξε ότι ο προστατευτής προστατευτισμό στα κράτη-μέλη και ιδίως στις κυβερνήσεις των κρατών μελών διαδραματίζει μεγάλο ρόλο και πρέπει να μας απασχολήσει αυτό το θέμα και να γίνουν προσπάθειες. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε έναν ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο και να μην έχουμε μία ενιαία οικονομική κυβέρνηση μου πήρατε τα λόγια από το στόμα και γι' αυτό πρέπει να προσπαθήσουμε να την υλοποιήσουμε. Ε, επίσης όσον αφορά τη συνθήκη της Λισαβόνας πιστεύω ότι ε, και αυτή η θεώρηση πρέπει να περιληφθεί στην έκθεσή σας διότι η ρόλη του κυρίου Βαν και της κυρίας ε, Άστον είναι επίσης σημαντική για να ε, ολοκληρώσουν το οικοδόμημα και τις διασυνδέσεις του και όσον αφορά το ρόλο του κυρίου Βαν Ρομπόη σαν επικεφαλής των κυβερνήσεων αν θέλετε να σας το πω ευθαρσός ο ρόλος αυτός πρέπει να αναλυθεί για να υπάρχει ένας ενιαίος κοινός χαρακτήρας

και με αυτό πρέπει να αναρωτηθούμε το, αυτό που είπατε κι εσείς. Δηλαδή τι εννοούμε με ορισμένα λόγια και πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν, υπάρχει στο θέμα της αγοράς πρόβλημα. Ε, για την αγορά κάθε κυβέρνηση θεωρεί ότι έχει τη δικιά της. Όλοι αναρωτιούνται τι είναι η αγορά, αναρωτιούνται αν θέλουν ενία ή κοινή αγορά αλλά ο χαρακτήρας του κοινού είναι πιο εύκολο να κατανοηθεί από τον πολίτη από το, ε, την ενία αγορά και γι' αυτό προτείνω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το κοινό αυτό χαρακτήρα ε, να τον διαχωρίσουμε και να ξανασκεφτούμε εάν θέλουμε να τονίζουμε την έννοια ενιαίο και θέλω να δώσω μια απάντηση και στην κυρία Κοράτσα γιατί νομίζω ότι εδώ με την έκθεση Γκρέχ ε, γίνεται ακριβώς το αντίθετο από αυτό που είπατε εσείς δηλαδή να υπάρχει μια εξειδανίκευση της ε, κοινωνικής αγοράς διότι έχουμε αποδείξει ότι η οικονομική πολιτική, η πολιτική των καταναλωτών και η κοινωνική πολιτική μπορούν να συνδυαστούν και κατά αυτόν τον τρόπο να υπάρξει κάτι θετικό για τις επιχειρήσεις και για τους πολίτες αν αντιμετωπίζονται όλα αυτά τα θέματα συλλογικά και συγκεράζονται. Και αυτό είναι το νέο στοιχείο στην πρόκληση που έχουμε αναλάβει και που προτείνει και σαν καινοτομία ο κύριος Μόντι ε, όσον αφορά την Ευρώπη. Εάν ακολουθήσουμε λοιπόν αυτή την σύνοδο πιστεύω ότι θα γίνουμε πιο αποδεκτοί από τους πολίτες ε, όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και την εσωτερική αγορά και αυτά ήταν τα σχόλια τα οποία ήθελα να κάνω. Ευχαριστώ. Κύριος Ροσφόρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στην πρώτη παρέμβαση όπως και άλλοι συνάδελφοι πήγαινα από τον ε, καθηγητή Γκρέσ προς τον καθηγητή Μόντι και τώρα κάνω την αντίστροφη πορεία ε, διότι η παρα τηρήσεις και των δύο είναι συμπληρωματικές και συγκλίνουν. Ξαναείπατε κύριε Μόντι πόσο σας ενδιαφέρει η ολιστική προσέγγιση και πρέπει αυτό να το ακολουθήσουμε μέχρι τέλους γιατί είναι ένας τρόπος για να δούμε με ένα νέο τρόπο τα πράγματα και κυρία Γκέπχαρντ εμένα δεν με ενοχλεί η έκθεση του κυρίου Γκρέχ να υπερβάλλει και να ξεπερνά το θέμα του καταναλωτή ε, δεν μπορεί κανείς να πει ότι δεν υπερομείνουμε τον καταναλωτή αλλά ε, πρέπει όχι μόνο να δείξουμε ε, μία σύγκληση προσεγγίσεων αλλά και μία σύγκληση των ρόλων των διαφόρων οικονομικών παραγόντων. Σήμερα το πριν λοιπόν δεν είπαμε γιατί αψηφά κανείς την ενία αγορά και μπορώ να σας πω ότι γίνεται στη χώρα μου που ισχύει όχι μόνο στη χώρα μου στα ιδρυτικά μέλη της ενώσεως και ίσως λιγότερο στα νέα ε, κράτη ε, διότι λέγεται ότι η ενιαία αγορά εντείνει τον ε, ανταγωνισμό δημιουργεί ανεργία διώχνει τις επιχειρήσεις που φεύγουν εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως άρα εμείς με την εσωτερική αγορά προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε την ανεργία αλλά αν δεν το διακηρύξουμε δεν γινόμαστε εμπιστευτοί. Πρέπει λοιπόν να προασπίσουμε τα δικαιώματα των καταναλωτών, να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη τους, να τους ε, ξαναδώσουμε τη σωστή θέση τους και όπως ελέγχθη για την ε, τηλεφωνία, για τις ε, υπηρεσίες τις τραπεζικές δόθη αντίθετη εντύπωση γιατί υπάρχουν ολιγοπόλια στο, στις υπηρεσίες τηλεφωνίας και στις τραπεζικές υπηρεσίες διότι ο, ο, ο πολίτης δεν μπορεί να επιλέξει το πακέτο που θα χρησιμοποιήσει μόλις βγει από τη χώρα του. Μπορούμε να ελέγξουμε την κατάσταση μόνο στη χώρα μας. Για να ενισχύσουμε λοιπόν την εσωτερική αγορά πρέπει να υπερβούμε τα όρια αυτά και να μην επιβεβαιώνουμε αυτά τα πολι ε, ολιγοπόλια όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος ε, Μόντι από τον προηγούμενο ρόλο του αλλά και να καταλάβουμε ότι οι καταναλωτές αφενός δεν καταλαβαίνουν ότι αγοράζουν πιο φθηνά αλλά ε, τον κοροϊδεύουν γιατί μειώνονται οι θέσεις εργασίας και σε ορισμένες αγορές δεν υπάρχει ουσιαστικός ανταγωνισμός αλλά συνεννόηση των ενδιαφερομένων. Αυτά είναι που πρέπει να καταλάβουμε καταπολεμήσουμε από κοινού. Και η σύγκληση μεταξύ των δύο θέσεων και συμφωνώ απολύτως με αυτά τα οποία είπε η κυρία Κοράτσα και άλλοι πρέπει να γίνει σε μία προβολή προς το μέλλον όπου νομίζω ότι η έρευνα για την ανάπτυξη και ε, για το περιβάλλον προχωρεί καλά και κάνω μία ερώτηση στον κύριο Μόντι είμαστε δέσμοι του χώρου που μπορούμε να κινηθούμε είμαστε μία από τις επιτροπές για την ανεργία εμείς δεν έχουμε ε, συνυπευθυνότητα για την καταπολέμηση της ανεργίας αλλά υπάρχει και μία παγίθευση ε, ξέρετε υπάρχει ε, ένας μεθυσμένος που ψάχνει τα κλειδιά του κάτω από ένα φως και δεν αντιλαμβάνεται ότι αν έχασε στα κλειδιά λίγο παραπέρα δεν θα τα βρει. Πρέπει λοιπόν και εμείς να απομακρυνθούμε από τις θέσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να ε, διευρύνουμε το πεδίο και να το πούμε και στον κύριο Μπαρόζο. Δηλαδή πέραν ε, της αναθέσεως έργου που σας έκανε ο κύριος Μπαρόζο πρέπει να απευθυνθούμε ε, σε όλους τους εμπλεκόμενους για να μπορέσει να ανακάμψει η εσωτερική εσωτερική Πολύ μ' άρεσε ε, ε, κύριο Μιλητά ε, το παράδειγμα με τα κλειδιά. Ε, θα ήθελα λοιπόν να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά υποθέτω ότι ο καθηγητής Μόντι θα θέλει να δευτερολογήσει. Καταρχήν η Επιτροπή αλλά έχουμε ε, ακόμη 20 λεπτά σύνολο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αντιπροσωπεύω εδώ την ε, Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς. Καταρχήν θα θέλω να κάνω ορισμένες παρατηρήσεις σχετικά με την έκθεση Γκρέχ και δεύτερον αναφερθώ στο που βρισκόμαστε όσον αφορά τις υπηρεσίες. Όσον αφορά την έκθεση συμφωνούμε στις γενικές γραμμές της εκθέσεως Γκρέχ γιατί εξετάζει την κατάσταση εσωτερικής αγοράς και τις δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζει. Οι περισσότερες από αυτές τις δυσκολίες αναφέρονται σε αυτή την έκθεση και ορισμένοι αναφέρθηκαν και σε άλλα θέματα και πιστεύω ότι ε, εάν είχαν προχωρήσει θα γνωρίζαμε επακριβώς τα της εσωτερικής αγοράς αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε ότι το βασικό πρόβλημα είναι ο συμβιβασμός της αγοράς με τους άλλους στόχους ε, της συνθήκης, δηλαδή κοινωνικούς, περιβαλλοντολογικούς στόχους οι οποίοι αναφέρθησαν και από την άποψή μας ο Επίτροπος Μπανιέ το είχε αναφέρει στην ακρόασή του στο Κοινοβούλιο. Δεν μιλάμε για την αποτελεσματικότητα της αγοράς σαν αυτό σκοπό, αλλά για να εξυπηρετηθεί ο πολίτης. Και πολύ σωστά είπε ο κύριος Ροσφόρ τώρα ότι ε, υπάρχουν συγκρούμενα συμφέροντα ε, υπάρχουν τα συμφέροντα του καταναλωτή που μπορεί να έχει καλές υπηρεσίες σε χαμηλή τιμή αλλά υπάρχουν ε, και οι ανεξάρτητοι οι ελεύθεροι επαγγελματίε οι εργαζόμενοι που θέλουν να προστατεύσουν τις θέσεις εργασίες τους υπάρχουν οι Ευρωπαίοι πολίτες και όλα αυτά τα θέματα ε, συγκρούονται στη λήψη των αποφάσεων και γι' αυτό αυτή τη στιγμή πρέπει να προσπαθήσουμε ε, να ρυθμίσουμε ε, και να συγκεράσουμε τα συμφέροντα για να εξυπηρετήσουμε τον πολίτη. Και αυτό το νέο έργο δεν είναι απλό. Πρέπει να προσπαθήσουμε η εσωτερική αγορά να ακολουθήσει τη στρατηγική 2020 και γι' αυτό πρέπει να προσπαθήσουμε να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερη αποτελεσματικότητα και στο σημείο αυτό θα πρέπει να ανταποκριθούμε. Από αυτή την άποψη λοιπόν πιστεύω ότι η έκθεση Γκρέκ καλύπτει αυτές τις απόψεις και όσον αφορά ε, τις ε, ε, προθεσμίες που ανέφερε ο κύριος Γκρέχ όσον αφορά τα, τις νομοθετικές επιπτώσεις για το 2011 μας μιλήσατε για ένα σύμφωνο εσωτερικής αγοράς και στην εσωτερική, στις υπηρεσίες μας το θέμα αυτό δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί και θα πρέπει να υιοθετηθεί σε επίπεδο Επιτροπής την επόμενη εβδομάδα και τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα γνωρίζει καλύτερα πώς θα προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Αλλά μόνο το 2011 περιμένουμε να προχωρήσουμε σε αυτό το θέμα και να έχουμε μία λευκή βίβλο ή και άλλα θέματα. Προς το παρόν μιλάμε για λευκή βίβλο η οποία είναι ανοιχτή και βεβαίως ε, ο στόχος δεν είναι μόνο να ληφθούν μέτρα όπου χρειάζονται αλλά και να υπάρξει ένα πάνελ δράσης για να ενημερώσουμε καλύτερα τους καταναλωτές και να ενισχύσουμε τη ε, σωστή εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου και γι' αυτό περιμένουμε τις προτάσεις του ε, καθηγητή Μόντι. Θα ήθελα να σας πω ότι όσον αφορά την Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να εντοπίσουμε τα, τους ελείποντες κρίκους στην αλυσίδα της εσωτερικής αγοράς εξετάζοντας συστηματικά πώς θα μπορέσουμε να συμβάλλουμε και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο τέλος Απριλίου θα αναλάβει τις αποφάσεις μας για να μπορέσει να τις συζητήσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τα σχόλια και για το χρονοδιάγραμμα. Σίγουρα η Επιτροπή θα θέλει να αντιδράσει στην ανακοίνωση και όντως δεν συμπεριλάβαμε τον όρο «χαμένος κρίκος» που είναι νέα ορολογία του Ευρώπη 2020. Τώρα κύριε Μόντι, μήπως θέλετε να εκφέρετε ορισμένες τελικές απόψεις. Θα είμαι πολύ σύντομος. Καταρχάς, σε σχέση με αυτά που είπε η κυρία Μπρόντερ αλλά και ο κύριος Κάρας για τον συντονισμό μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης 2020 και του δικού μου έργου όσον αφορά την εσωτερική αγορά. Πιστεύω ότι στο τέλος θα καταλήξουμε σε αρκετά ορατή συνόχη. Εγώ στην έκθεσή μου συνεργάζομαι στενά με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ ΜΑΡΚΤ αλλά και με τον Επίτροπο κύριο Μπαρνιέ σε πολιτικό επίπεδο και η μικρή ομάδα μου που ασχολείται με την έκθεση βρίσκεται, εδρεύει στη γραμματεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ασχολείται, βρίσκεται στον πυρήνα της επεξεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2020. Και όλα αυτά νομίζω ότι θα οδηγήσουν σε πολύ ορατή συνοχή. Να πω επίσης ότι συμφωνώ με αυτά που είπαν με διαφορετικούς τρόπους οι κύριοι Κάρας και Ροσφόρ ότι θα υπάρξουν ε, θέματα που είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών, είτε καθενός ξεχωριστά, είτε όλων μαζί, για αρμοδιότητες που είναι περισσότερο διακυβερνήτικες παρά κοινοτικές. Και σίγουρα στην έκθεσή μας θα κάνουμε κάποιες συστάσεις προς ε, το όργανο που ζήτησε την έκθεσή μας, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά αν χρειαστεί και για το Συμβούλιο και αν μπορώ να τολμώ να το πω και για το Κοινοβούλιο και βεβαίως τα κράτη-μέλη. Τώρα όσον αφορά τη σχέση μεταξύ αγοράς και κοινωνικής διάστασης. Να υπογραμμίσω καταρχάς, ε, κύριε Ράπτη, ότι όντως είχα διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους. Αναφέρθηκα γενικά στα ενδιαφερόμενα μέρη, αλλά είχα πολύ νωρίς διαβουλεύσεις με το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων, τη Business Europe και άλλες ε, επιχειρηματικές ενώσεις, ενώ επίσης την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει και μια τελική συνεισφορά των κοινωνικών εταίρων στην έκθεσή μου, μια κοινή συνεδρίαση Ευρωπαϊκής Συνοσπονδίας Συνδικάτων και Business Europe. Επίσης, θα ήθελα να συμφωνήσω με αυτό που είπε η κυρία Κοράτσα Μπίλτ ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να σταθούμε στο ύψος μας για τον διεθνή παγκόσμιο ανταγωνισμό. Όντως αυτό θέλουμε να κάνουμε στα πλαίσια της εσωτερικής αγοράς. Εγώ βεβαίως δεν θα προτείνω, δεν είναι δική μου αρμοδιότητα, δεν θα προτείνω λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να αυξήσει το περιεχόμενο, το βάρος, το κόστος των κοινωνικών πολιτικών της. Αυτό δεν είναι δικό μου θέμα. Αυτό που είναι δικό μου θέμα είναι οι τομείς οι οποίοι σε επίπεδο εντυπώσεων επηρεάζουν τους πολίτες προκειμένου οι πολίτες να μπορούν να διαπιστώσουν στην πραγματικότητα ή όπως το καταλαβαίνουν ότι η εσωτερική αγορά επιτρέπει στα κράτη-μέλη να ενδυναμώσει την κοινωνική προστασία. Γιατί αν δεν γίνεται αυτό, τότε έτσι ακριβώς είναι που δημιουργούνται εχθροί για την Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ των πολιτών. Και αυτό θα το αναφέρω σαφώς στην έκθεση. Τέλος, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ρωτήσω εσάς και τον εισηγητή, τον κύριο Γκρέκ, αν είναι δυνατόν να βρισκόμαστε σε στενή επαφή τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες, γιατί νομίζω ότι θα αυτό θα είναι προς το συμφέρον του δικού μου έργου, αλλά και προς το κοινό μας συμφέρον. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε ενδελεχώς ε, το χρονοδιάγραμμά μας και γενικά τις συνεργίες και τους άλλους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να συνεργαστούμε προκειμένου να επιτύχουμε αυτή την ολιστική προσέγγιση για την εσωτερική αγορά. Ευχαριστώ. Ναι, το εξετάζουμε αυτό και τώρα μόλις που μιλούσατε κοιτάζαμε το χρονοδιάγραμμα. Όσον αφορά τώρα τις τροπολογίες για τους συναδέλφους Νομίζω ότι ο κρίσιμος μήνας για τις συζητήσεις θα είναι ο Μάιος. Η κυρία Μπρόντ μας μίλησε και για ενδεχομένως πιο φιλόδοξες προτάσεις, ίσως κάποια λευκή βίβλο. Το σημαντικό λοιπόν είναι ψηφοφορία για την έκθεση Γκρέχ μέχρι τις 28 Απριλίου στην Επιτροπή προκειμένου να μπει στην Ολομέλεια της 19ης Μαΐου. Σας υπενθυμίζω ότι 25-26 Μαΐου είναι το Συμβούλιο Ανάπτυξης ενώ η έκθεση Μόντι αναμένεται για τα τέλη Απριλίου και η, έκθεση της, η ανακοίνωση της Επιτρόπου μέσα Μαΐου. Άρα λοιπόν πρέπει να έχουμε ψηφίσει την έκθεση Γκρέχ μέχρι τον Ιούνιο. Διαφορετικά έχουμε χάσει το στίχημα. Νομίζω ότι επειδή έχουν γίνει πολλές διαβουλεύσεις από τον κύριο Γκρέχα, έχουμε μια καλή πρόταση αυτή τη στιγμή. Σας προτείνω λοιπόν 13 Απριλίου 6 το απόγευμα προθεσμία για τις τροπολογίες, λίγο στενό το όριο, αλλά έχετε μέχρι την επόμενη εβδομάδα να καταθέσετε τροπολογίες προκειμένου να μπορέσουμε να ψηφίσουμε την έκθεση στις 28 Απριλίου, ενδεχομένως ε, και με κάποιες συμβιβαστικές τροπολογίες, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι θα περάσει το θέμα στην Ολομέλεια του Μαΐου. Και μετά ανεξάρτητα από το τι θα κάνει η Κομισιόν θα μπορέσουμε εμείς να έχουμε μια καλή έκθεση που θα στείλουμε και στο Συμβούλιο και στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας. Εξαιρετικά κύριε Πρόεδρε. Απλά δώστε μου 30 δευτερόλεπτα γιατί ξέχασα ένα πολύ σημαντικό θέμα που έθεσε η κυρία Γκέπχαρτ στην δεύτερη παρέμβασή της όσον αφορά την οικονομική διακυβέρνηση. Από την πλευρά μου θα προσπαθήσω να σας εξηγήσω όσο πιο σαφές γίνεται την σχέση μεταξύ της ανάπτυξης της εσωτερικής αγοράς και αυτής της νέας προθυμίας να αποκτήσουμε οικονομική διακυβέρνηση. Και να πω ότι όσες περισσότερες προσπάθειες κάνει το Κοινοβούλιο για να φανεί αυτό, ο σύνδεσμος, αυτή η σχέση, τόσο καλύτερα για αυτήν το πραγματικό ενιαίο κόσμο της εσωτερικής αγοράς. Και αυτό ισχύει και για την οικονομική διακυβέρνηση. Λούι, νομίζω ότι έτυχε πολύ θετική υποδοχή η έκθεση. Συγγνώμη, εκ μέρους του ΕΛΚ να ρωτήσω αν μπορούμε να αναβάλουμε την ε, προθεσμία μέχρι το τέλος της εβδομάδας τότε δεν θα έχουμε μεταφράσει όλες τις γλώσσες για την ψηφοφορία στις 28 Απριλίου. Μας πιέζει ο χρόνος δυστυχώς. Νομίζω ότι είναι υπερβολικά σύντομος ο χρόνος. Αυτή είναι η θέση του ΕΛΚ, κύριε Πρόεδρε. Το πρόβλημα είναι ότι δεν θα έχουμε τις τροπολογίες σε όλες τις γλώσσες για ψηφοφορία στις 27 Απριλίου και αν καθυστερήσει η ψηφοφορία μετά τις 28 Απριλίου δεν θα μπορέσουμε να ψηφίσουμε την έκθεση στην Ολομέλεια το Μάιο που είναι η σημαντική ημερομηνία. Η μόνη άλλη επιλογή είναι να μην έχουμε τροπολογία σε όλες τις γλώσσες και αυτό είναι πολύ ευαίσθητο θέμα για κάποιους συναδέλφους. Ας το θέσω αλλιώς. Θα ζητήσω από τη Γραμματεία να εξετάσει το θέμα. Αν η άποψη της Επιτροπής είναι ότι πρέπει να είναι έτοιμη η έκθεση για το Συμβούλιο, η Γραμματεία θα έρθει σε επαφή με τις μεταφραστικές υπηρεσίες και θα μπορούσαμε ίσως να έχουμε ένα πυρήνα γλωσσών οι οποίες θα επαρκούν. Θα προσπαθήσουμε να σας δώσουμε τουλάχιστον μία μέρα χρόνο μέχρι την Τετάρτη. Συμφωνούμε επί της Τετάρτης 14 του μηνός και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Δώδεκα το μεσημέρι, Τετάρτη 14 Απριλίου. Έχετε όλο το βράδυ της Τρίτης για να τις εξετάσετε. Ο Λουί Γκρέκ τώρα παρακαλώ. Πραγματικά θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους παρενέβησαν, σκιώδεις, εισηγητές, συντονιστές, όλους τους. Είναι πραγματική πρόκληση αυτού του input και αυτό είναι πραγματικά η ιδέα που μας ενέπνεε. Αυτό το οποίο απορρέει από τη συζήτηση είναι ότι η εσωτερική αγορά χρειάζεται πραγματικά κάποιον ηγέτη ηγετικό ρόλο για να, να διαφύγει από τις συμπληγάδες και με τη γνώση του ο κύριος Μόντι και τις ιδέες του μπορεί να παράσχει αυτή την ηγετική ιδιότητα από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ηγετικό ρόλο για να προχωρήσει η εσωτερική αγορά πιο αποτελεσματικά. Ένα σημείο που αναφέρθηκε είναι ότι δεν κάλυψα κάποιους τομείς. Πρώτον, η γραμματεία μου έλεγε ότι δεν θα έπρεπε μια και 20.000 ψηφία επιτρεπόντουσαν ως εύρος της έκθεσης δεν μπορούσα όλα να τα συμπεριλάβω. Δεύτερον, νομίζω ότι σε σχέση με το στόχο την επίτευξη του, της εσωτερική εσωτερικής αγοράς για τους πολίτες και καταναλωτές έπρεπε να έχω μια πειθαρχημένη ε, έκθεση με προτεραιότητες. Διαφορετικά είναι τόσο τεράστια η εμβέλεια αυτής, ε, αυτού του θέματος και πνευματικά δικαιώματα και ιδιοκτησία και τόσα πολλά άλλα θέματα μπορούν να καλυφθούν από την έκθεση αν όπως είχα ακολουθήσει την πορεία της ευρύτερης έκθεσης αυτό θα ήταν αντιπαραγωγικό. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν πρόκειται εδώ για ένα ευχολόγιο, μια ατζέντα που θα θέτει επί παντός του επιστητού ε, ρόλο προτεραιότητας. Δεν μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Θα έπρεπε τα ουσιοδέστερα να επιλεγούν. Η επικέντρωση να είναι η εστίαση στους πολίτες και καταναλωτές. Να είναι στο τι πραγματικά μπορεί να αναζωογονήσει και πρέπει να αναζωογονήσει την εσωτερική αγορά. Ακριβώς αυτό το σταυροδρόμι της εσωτερικής αγοράς. Υπάρχει μεγάλη ευκαιρία να υπάρχει όχι ολοκλήρωση αλλά κατακαιρματισμός ε, της ε, εσωτερικής αγοράς. Πρέπει να θέσουμε προτεραιότητες. Δεν μπορούμε να είμαστε υπερβολικά στον φόδης. Καλύτερο θα είναι να είμαστε συνετοί, σόφρονες και αυτή την επιλογή ακολούθησα, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Ευρώπη, πιστεύω να έχει μια εσωτερική αγορά που πραγματικά θα την εκτιμούν οι πολίτες και θα εκφράζουν εμπιστοσύνη σε αυτήν ως καταναλωτές. Είπα ολιστική, σφαιρική, συνολική δηλαδή προσέγγιση στην έκθεσή μου. Έχουμε αυτούς τους τέσσερις άξονες, αλλά έχουμε ένα πέντα, πέμπτο άξονα που χρειαζόμαστε. Δηλαδή τον πολίτη και τον καταναλωτή ως πέμπτο άξονα. Είναι ευρύτατο το, ε, το πλαίσιο και είναι ένα νέο πρότυπο νοτροπίας και ε, σκέψης ε, ως προσέγγισης. Όχι μόνο οι πολίτες και οι καταναλωτές αλλά και το γεγονός ότι πρέπει να υπάρχει αναφορά συγκεκριμένη, ισχυρή στην έκθεσή μου. Πρέπει να εξετάσουμε και να δούμε πώς θα μπορέσει να λειτουργήσει αποτελεσματικά η εσωτερική αγορά. Ξεπερνά ιδεολογικά εσκαμμένα και πλαίσια ε, και διαχωριστικές γραμμές αυτή η έκθεση. Δεν πρέπει να είμαστε ε, σε διαχωρισμένα πλαίσια. Πρέπει να λειτουργήσει η εσωτερική αγορά. Αυτό είναι η αποτελεσματική επικέντρωση, η κέρια επικέντρωση. Και αυτό που προτείνω ως deliverables που πρέπει να επιτευχθούν δηλαδή ως αποτελέσματα ε, βλέποντας ε, τι μπορεί να επιτευχθεί. Κάτι συγκεκριμένο πρέπει να γίνει, αυτό θέλω να γίνει δεν ε, ε, έχω μεγάλη πίστη σε πολλά συνθήματα και πολλές ε, διαφορετικές έννοιες. Θα ήθελα να έχουμε μια αποτελεσματική δράση που θα επιτελέσει στόχους αποτελεσματικά. Κάτι που θα μεταφράζει την εσωτερική αγορά με αποτελεσματικό εποφελή τρόπο σε όλους, για όλους τους εμπλεκόμενους. Τις επιχειρήσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εταιρείε, αλλά πολύ περισσότερο για τους ίδιους πολίτες και καταναλωτές κυρίως. Σας ευχαριστώ πολύ λέει ο Πρόεδρος, για την ανακεφαλαίωση. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέφους για τις πολύ καλές ε, παρεμβάσεις και συνεισφορές τους. Ήταν μια πραγματικά καλή ευκαιρία να έχουμε μια τόσο εκτενή συζήτηση. Ευχαριστώ ιδιαίτερα εσάς καθηγήτα Μόντι για το ότι ήρθατε εδώ στην Επιτροπή μας και με μεγάλη χαρά θα σας προσκαλέσουμε για να παρουσιάσετε την τελική σας έκθεση την οποία δημονούμε να δούμε και τώρα λίγη συνεδρίαση. Απλά θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής μας θα είναι στις 27 και 28 Απριλίου. Επόμενη συνεδρίασή μας εδώ στις Βρυξέλλες. Θα ψηφίσουμε στις 10 η ώρα το πρωί έχοντας και ε, ψήφιση της έκθεσης GREC θέλω να σας ενημερώσω την Δευτέρα της επόμενης εβδομάδας η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς θα έχει ένα workshop για τις αλλαγές όσον αφορά το, τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας και τις υπηρεσίες σχετικά έχουμε συζητήσει και με την Οικονομική Επιτροπή για το πώς μπορούμε να υπάρξει ένα input σε σχέση με τους καταναλωτές. Προσκαλείστε να συμμετάσχετε σε αυτό το workshop στις Βρυξέλλες το απόγευμα της επόμενης Δευτέρας στις 3 το απόγευμα. Σας ευχαριστώ όλους σας και προσβλέπω να σας ξαναδώ κατά τέλη Απριλίου. Γεια σας.